Okay, friends, we'll start the... Αγαπητοί φίλοι, να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Με ιδιαίτερη χαρά δεχόμαστε εδώ τον, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για πολλά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. προετοιμασία του επόμενου προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και πιο συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι η χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να τον ρωτήσετε για πολλά και διαφορετικά ζητήματα και εκείνο σίγουρα θα προσπαθήσει να απαντήσει όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Κύριε Κατάινεν, έχετε το λόγο για μια εισαγωγή σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και όλους τους ευρωβουλευτές που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να συζητήσω μαζί σας όλα αυτά τα θέματα. Ναι, θα πω δύο λόγια, πρώτα απ' όλα για τις δεξιοτεχνίες και συνέχεια θα αναφερθώ στο επενδυτικό πρόγραμμα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μετά θα μιλήσω για την χαλιβουργία και τέλος για τον κοινωνικό διάλογο και τα κοινωνικά δικαιώματα. Για τις δεξιοτεχνίες πρώτα απ' όλα. Ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να δημιουργήσει μια τέτοια ατζέντα στόχους δηλαδή για τις δεξιοτεχνίες είναι γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα δυστυχώς καταλαβαίνουμε και εγώ το πιστεύω αυτό ότι η δεξιοτεχνία η κατάρτιση δεν βρίσκεται πάνω πάνω στην πολιτική ατζέντα όσο θα έπρεπε. Και είναι κρίμα. Όλοι έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε για την ε, μεταβιομηχανική επανάσταση, για τις ε, αλλαγές, ε, πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τους εργαζόμενους όσον αφορά τα προσόντα, γιατί αλλάζουν αυτά. Και πολλές φορές οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν έχουν αρκετά προσόντα και δεξιοτεχνίες για να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της απασχόλησης, πόσο μάλλον στις μελλοντικέ. Γι' αυτό λοιπόν, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πολλές εξουσίες επί του θέματος, θελήσαμε να επικεντρωθούμε στο θέμα των δεξιοτεχνιών. Διαφέρουν μεταξύ χωρών μελών κατά πολύ. Γενικά ε, μιλώντας έχουμε εντοπίσει κάποια ζητήματα στα οποία θα έπρεπε να δώσουν περισσότερη προσοχή οι χώρες μέλη και να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Σε μερικές χώρες υπάρχει περιθώριο ε, ελιγμών για να υπάρξει καλύτερη κατάρτιση. Σε άλλες χώρες είναι τα θέματα της ε, εκπαίδευσης, της μάθησης ακόμα και στις περισσότερες χώρες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των μεταναστών. Είναι περιττόν να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν ε, οι γνώσεις, οι δεξιοτεχνίες και τα προσόντα στην Επιτροπή αυτή εδώ που βρισκόμαστε. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά θα σας δώσω κάποια νούμερα. Σήμερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όσον αφορά τους ενήλικες και τις ε, δεξιοτεχνίες τους. Έχουμε πάνω από 70 εκατομμύρια οι οποίοι δεν έχουν αρκετά κατάλληλα προσόδια και δεξιοτεχνίες. 25% των ε, ενηλίκων δεν έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και πάρα πολλοί δουλεύουν ε, σε δουλειές που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους οι γυναίκες είναι το 60% και σίγουρα η μόρφωσή τους είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Το 40% των επιχειρήσεων από την άλλη μεριά δεν βρίσκουν ανθρώπους με τα προσόντα που χρειάζονται και πολύ λίγοι διαθέτουν επιχειρηματικά προσόντα για να δημιουργήσουν τη δικιά τους την επιχείρηση. Όλες αυτές οι ικανότητες λοιπόν δεν έχουν αποτελέσει την προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντα στις χώρες μέλη. Θα έπρεπε όμως. Επιπλέον, στην εποχή των ψηφιακών αλλαγών, η Ευρώπη δεν διαθέτει ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα. Άρα λοιπόν την ε, κατάρτιση σε αυτούς του τομείς πρέπει να τη δούμε σαν προτεραιότητα και να γίνουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των χωρών μελών. Η Επίτροπος Τάισον στις 7 Ιουνίου τα παρουσίασε στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για την εγγύηση ικανοτήτων και προσόντων υποσχόμενη βοήθεια στις χώρες μέλη ώστε οι άνθρωποι που δεν έχουν ευκαιρίες να καταρτιστούν καλύτερα να μπορέσουν να το κάνουν. Επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για ε, τις δεξιοτεχνίες, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε δεξιοτεχνίες και προσόντα καλύτερα μεταξύ των χωρών μελών. Και τρίτον, προωθούμε και την συνεργασία όσον αφορά το θέμα της δεξιοτεχνίας σε διάφορους τομείς, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να εντοπίσουν τα προσόντα που χρειάζονται και να εντοπίσουν και λύσεις για να τα βρούνε. Έπειτα, για την αγορά εργασίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους υπηκόους τρίτων χωρών. Σίγουρα χρειάζεται ένα νήμα που να συνδέει την εκπαίδευση με την ε, μόρφωση, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, κατάρτιση και απασχόληση. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και ένα πουλ δεξιοτεχνήτων, φροντίζοντας για όλα τα επίπεδα. Προκειμένου τώρα να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη για να υλοποιήσουν τις προτάσεις που κάνουμε για το διάστημα από το 2014 μέχρι το 2020, πάνω από 27 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για αυτό το σκοπό. Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και θέλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό. Θα σας πω και δύο λόγια τώρα για το επενδυτικό σχέδιο. Θα ξεκινήσω από τον τρίτο πυλώνα, γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού προγράμματος. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή έχει αναλύσει την οικονομική κατάσταση έχει λάβει υπόψη της και την κοινωνική προοπτική και τις δεξιοτεχνίες στις χώρες μέλη. Έχουμε εντοπίσει τα μεγαλύτερα εμπόδια, κυρίως στις χώρες μέλη, όσον αφορά τις επενδύσεις, γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Ε, του χρόνου λοιπόν στις συστάσεις μας θα συμπεριλάβουμε συστάσεις που να, επικεντρώνονται σε αυτά τα εμπόδια για τις επενδύσεις. Γιατί θέλουμε να θαρρύνουμε τις χώρες μέλη να καταργήσουν τα εμπόδια αυτά και έτσι να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να αυξηθεί η απασχόληση συνεπώς. Εντοπίσαμε επίσης και αυτό που λέω ευρωπαϊκά μόνο εμπόδια. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα ποια είναι αυτά. Συζητούμε με την Eurostat προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουν τις χώρες μέλη και κυρίως τους επενδυτές, γιατί υπάρχουν ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα επενδύσεις κοινές, για να δούμε τι θα συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος και τι όχι. Οι επενδυτέ τη χρειάζονται αυτή τη βοήθεια και ακόμα περισσότερο επειδή τα επιχειρηματικά μοντέλα αλλάζουν. Πολλά τέτοια ε, σχέδια δημοσίου τομέα έχουν διαφορετική μορφή από ό,τι είχαν κατά το παρελθόν. Ένα άλλο παράδειγμα των εμποδίων από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πώς θα συνδυάσουμε το ΕΦΣΥ, το επενδυτικό αυτό ταμείο, με τα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε δώσει λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές και τώρα βοηθούμε τις χώρες μέλη για να εκπονήσουν προγράμματα και να μπορέσουν έτσι να επωφεληθούν. Και τέλος, υπάρχουν και ευρωπαϊκές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει ότι πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο στην εσωτερική αγορά. Γνωρίζετε την, το εμβληματικό μας ε, σχέδιο για την ε, Ένωση κεφαλαίων. Ξέρετε ότι περιλαμβάνουμε και σχέδια για τις μεταφορές και λοιπόν όλα αυτά είναι σχέδια που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά και που θα επηρεάσουν κατά πολύ θετικά το επενδυτικό κλίμα. Θα αναφερθώ τώρα πιο συγκεκριμένα στο ΕΦΣΙ, στο επενδυτικό ταμείο. Προς το παρόν πάει καλά. Θα σας δώσω κάποια νούμερα. Θα τα βρείτε όλα στο διαδίκτυο. Και αν κάποιος ε, δεν με παρακολουθεί στο Twitter, ε, ας με παρακολουθήσει γιατί και εκεί τα βάζω. Λοιπόν, το ΕΦΣΥ έχει στηρίξει προγράμματα και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τραπεζών, αλλά και σε επίπεδο υποδομών με 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένουμε έτσι να έχουμε επενδύσεις επιπλέον της τάξης των 107 δις. ...185 ε, συμφωνίες έχουμε ανάμεσα στο ΕΦΣΙ και μεσαίες τράπεζες και αυτές οι 185 συμφωνίες θα οδηγήσουν σε χρηματοδότηση 248.000 ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, έχουμε τρεις τράπεζες οι οποίες έχουν προχωρήσει σε τέτοια συμφωνία και βοηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ιταλία 28 τράπεζες που θα βοηθήσουν 44.000 Ιταλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση. Βλέπετε λοιπόν ότι όντω πρόκειται για επένδυση αφού βοηθάμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε και 78 ε, άλλα επενδυτικά σχέδια, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε παρετέρω επενδύσεις. ...27% για την ενέργεια, 25% για τις μικρομεσαίες, ψηφιακά 12% μεταφορές 6%, κοινωνικές επενδύσεις 3%. Το πιο σημαντικό βέβαια στοιχείο είναι ότι 80% των 107 δισεκατομμυρίων έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα οι δημόσιες επενδύσεις ε, οδηγούν σε ιδιωτικές επενδύσεις με τη σειρά τους. Πολύ έχουν πει εδώ ότι δεν πρόκειται για φρέσκο χρήμα, ότι το ΕΦΣΙ δεν ε, δίνει κατευθείαν χρήματα. Δίνει όμως γιατί πρόκειται για χρήματα τα οποία έρχονται στην αγορά. Χαλιβουργία τώρα. Θα σας πω ποια είναι η κατάσταση στην αγορά αυτή. Το Μάρτιο εγκρίναμε την ε, ανακοίνωσή μας για βιώσιμη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Βασιζόμαστε σε πέντε πυλώνες. Επιτάχυνση της έγκρισης μέτρων αντι-dumping. Ε, ενισχύοντας την παγκόσμια δυνατότητα, καινοτομία, δεξιοτεχνίες, ε, επικέντρωση σε πολιτικές όπως είναι ο ανταγωνισμός, η ενέργεια και η κυκλική οικονομία. Στηρίζουμε συνολικά τον κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, επανεισάγει σύστημα που έχει να κάνει με την τιμολόγηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε λοιπόν το dumping στην Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε έρευνες όσον αφορά το φαινόμενο αυτό. Εμπορικά μέσα τώρα και αυτά θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του κλάδου. Πάντως, ο κύριος στόχος μας είναι βιώσιμες λύσεις ώστε τα προβλήματα ικανότητας του κλάδου να αντιμετωπιστούν. Και διμερός κάθε φορά και πολυμερός. Διμερός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πολλαπλασιάσει τις επαφές της με τους κύριους ε, παραγωγούς και με την Κίνα γιατί πήγα στην Κίνα πριν από ένα μήνα για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα με τον Αντιπρόεδρο. Και σε επίπεδο όσα επίσης συζητιώνται αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι εξότιμοι ευρωβουλευτές, θα ολοκληρώσω αναφερόμενο στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κοινωνικά δικαιώματα, τον κοινωνικό πυλώνα. Δεδομένων των όσων πετύχαμε μέχρι τώρα, έχουμε τη σύσταση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της μακροχρόνιας ανεργίας. Με σκληρή δουλειά καταφέραμε να πετύχουμε διαπραγματεύσεις για μια πλατφόρμα όσον αφορά την αδήλωτη εργασία και να μεταρρυθμίσουμε το χάρτη για το δίκτυο απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενισχύσει επίσης και τις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορους τομείς ήρθε σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά τις μελλοντικέ προκλήσεις για μετά το 2016 αλλά και όσον αφορά τις αναχώρα εκθέσεις και τις αναχώρα συστάσεις. Στην απασχόληση και τις κοινωνικές ε, υποθέσεις έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους βάσει του άρθρου 154 για τις διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους και όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Θα συνεχίσουμε με τον κοινωνικό διάλογο γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι θα πετύχουμε μόνο με τον κοινωνικό διάλογο. Αυτός παίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια και το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση που μπορεί να βοηθήσει πολύ να ανακουφιστούν απολυμένοι εργαζόμενοι. Η ατζέντα επίσης για τις νέες δεξιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μπορεί να βοηθήσει στην ισορροπία μεταξύ και προσφοράς με πειραματικά προγράμματα όπως είναι αυτό για την όθηση των δεξιοτεχνιών και άλλα μεταξύ άλλων και στον τομέα της χαλιβουργίας. Και τέλος, 8 Μαρτίου φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι για τον Ευρωπαϊκό Πυλόν όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης. Έφτασε η στιγμή να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση μέσα στα πλαίσια της νέας οικονομίας και της νέας κοινωνίας που βέβαια επηρεάζεται και από την ελευθέρωση αλλά και την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο οι κοινωνικές μας πολιτικές στηρίζουν πραγματικά τους πολίτες και κατά πόσο τους προστατεύουν από κινδύνους. Μπορούν, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την αγορά εργασίας ή είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Θα περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική μας οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Ποιοι από σας θα ήθελα να θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσω με τους συντονιστές. Ο κ. Κάζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Άντι Πρόεδρε που είστε εδώ μετά το γεύμα για να μας κάνετε την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις βασικά. Νομίζω ότι το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να διασφαλίσουμε επενδύσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Οι επενδύσεις όμως, οι οποίες όταν δεν συνοδεύονται από διαφορετικές αλλαγές, δεν έρχονται. Απαιτούνται λοιπόν πολιτικές αποφάσεις με σωστό προγραμματισμό, εφαρμογή αυτών των αποφάσεων και προπαρασκευαστική δουλειά συμβουλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προώθησης των μικρομεσαίων είναι απαραίτητες. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες. Και δεύτερον, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, μπορείτε να μας αξιολογήσετε λίγο τι έγινε με τον πρώτο χρόνο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του σχεδίου Juncker δηλαδή. Βελτιώνεται η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίνσκι. Thank you, Madam was not aware that I was still... Δεν ήξερα ότι μετά από τη συνάντηση των συντονιστών το πρωί θα έπαιζε αυτό το ρόλο σήμερα το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Αντιπρόεδρε, το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε βρίσκεται στο κέντρο των ανησυχιών, αν θέλετε, της Επιτροπής μας. Απασχόληση, κατάρτιση είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση των επενδύσεων με τις μεταρρυθμίσεις και την επίτευξη κάποιων στόχων που είναι αν θέλετε βασικά η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας. Αναφερθήκατε στη σημασία που έχει η ποιότητα των ικανοτήτων και των γνώσεων. Αναφερθήκατε επίσης και στις ψηφιακές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για τους εργαζομένους. Όλα αυτά τα οποία είπατε και κάποια άλλα θέματα που γνωρίζουμε συνδέονται πολύ με την αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανισότητα έχει και μια εδαφική διάσταση και έχει σχέση με την έλλειψη γνώσεων σε περιοχές σε στασιμότητα οικονομική, σε περιοχές με ισχυρό περιφερειακό χαρακτήρα και υπάρχουν και περιοχές τις οποίες οι ευκαιρίες είναι περισσότερες ε, και όπου παρατηρούνται όμως κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Στα πλαίσια της παρουσίασής σας, στην ουσία εσείς δεν αναφερθήκατε καθόλου στο θέμα της συνοχής και νομίζω η συνοχή είναι κεντρικό θέμα εδώ. Νομίζω ότι και ο κύριος Κάζα θέλησε να το θέσει αυτό. Οι επενδύσεις φυσικά από μόνες τους δεν φτάνουν. Φυσικά είναι απαραίτητες αλλά δεν φτάνουν. Θα πρέπει να δούμε οι επενδύσεις αυτής αυτές τι κατεύθυνση έχουν, τι αποτελέσματα δίνουν και σε ποιο βαθμό βοηθούν την μεγαλύτερη συνοχή στην κοινότητα. Και τώρα να αναφερθώ σε κάποια μικρότερα επιμέρους θέματα, τα οποία με απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό. Πρώτον, η ανακοίνωση της Επιτροπής το Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τη συνεισφορά των διαφθρωτικών ταμείων στο στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων που και στις λεγόμενες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή καταρχάς δεν νομίζω ότι εκπληρεί τις απαιτήσει ε, της παραγράφου 3 του CPR που ζητά να υπάρξει έκθεση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι απλή ανακοίνωση. Δημιουργία των ε, λειτουργικών προγραμμάτων, ε, ειδικά χαρακτηριστικά μεμονωμένων χωρών μελών, υπάρχει ανάγκη από αναλυτικές παρουσιάσεις και έτσι θα καταλήξουμε στα κατάλληλα συμπεράσματα. Συν της άλλης, πέρα από τον ελλειπτικό χαρακτήρα της παρουσίασής σας, υπήρξε και καθυστέρηση στην έκδοσή της. Για την επόμενη περίοδο λοιπόν πώς θα διορθώσετε κάπως τα πράγματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι έκανε μέχρι τώρα καλά τη δουλειά της με την ανακοίνωση αυτή ή θα μας παρουσιάσει την επόμενη φορά μια πραγματική ανάλυση των ευρημάτων της. Χάρη στις προσπάθειες που έκαναν οι συνεργάτες μου, είδαμε ότι γίνεται δουλειά σε επιμέρους επίπεδο, γίνεται δουλειά σε τομεακό επίπεδο και θα πρέπει να είναι ενημερωμένο το Κοινοβούλιο για να συμμετέχει σε μια σοβαρή συζήτηση. Ένα άλλο θέμα. Εδώ είχαμε πριν μερικές μέρες ε, μία παρουσίαση του προγράμματος στήριξης των διαφθρωτικών αλλαγών, το οποίο φαίνεται ότι προχωρά και αυτή η πρόθεσή σας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επενδύσεων, το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς την κατεύθυνση αυτή. Στην ανακοίνωση που έκαναν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακούστηκε, είπαν ότι τα χρήματα αυτά βγαίνουν από κάποια τμήματα της τεχνικής βοήθειας από τη συνοχή δηλαδή και μπαίνουν στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αυτό λιγάκι περίεργο μας φαίνεται, μας το να παίρνετε δηλαδή από τη διαδικασία της συνοχής και να τα βάζετε στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και αυτό αφορά και εμάς και την Επιτροπή ε, ε Μεταφορών και υπονομεύει τις προσπάθειες, αν θέλετε, συνοχής οι οποίες γίνονται και στα πλαίσια του εξαμήνου και προβλέπονται από τη συνθήκη. Υπάρχουν ερωτηματικά λοιπόν γύρω από αυτά τα οποία κάνετε. Και η απάντηση που μας είχε δώσει στην αρχική μας ερώτηση εδώ και δύο μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορεί να δώσει εξηγήσεις δηλαδή για τη μεταφορά των πιστώσεων αυτών και τη χρησιμοποίησή τους σε προγράμματα τα οποία δεν συνδέονται με τους στόχους της συνοχής παρά μόνον δευτέρευόντους. Υπάρχουν ερωτηματικά για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει εις πέρα στην αποστολή της, εκτελεί αν θέλετε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται και το στρατηγικό πρόγραμμα μέχρι τώρα. Σύμφωνα με γνωστά δεδομένα και ακούστηκε αυτό και στην Ολομέλεια και σε συναντήσεις σαν τη δική μας δόθηκαν στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμα πείσει ότι υπάρχει ε, αυτή η πετυχημένη διαδικασία αν θέλετε προσέλκυσης επενδύσεων που δεν θα υπήρχαν κατά τα άλλα αν δεν υπήρχε το στρατηγικό πρόβλημα, πρόγραμμα για όλα αυτά τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε, τα 78 μίζωνα προγράμματα επενδύσεων. και σε ποιο βαθμό τα προγράμματα αυτά συνεισφέρουν και με τη σειρά τους στη συνοχή ή μήπως ε, εκεί σταματά αν θέλετε η δράση τους και ίσως να αναμείνουμε στο μέλλον και μια αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τώρα μακρηγορώ λιγάκι. Έχω αναφέρει πάρα πολλά θέματα, είναι αλήθεια. Μία τελευταία ερώτηση. Αυτές τις ανησυχίες τις οποίες έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο και σε επίπεδο ολομέλειας και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών καλύπτονται από τη δράση σας. Ή μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και λυπάμαι που το λέω αυτό, το μόνο που κάνει είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης ουσιαστικά, μια εκστρατεία πληροφόρησης. Και αυτό δημιουργεί μια κάποια δυσφορία, μια κάποια δυσθυμία στον τρόπο με τον οποίο προσελκύονται οι επενδύσεις και στον τρόπο με τον οποίο έρχονται οι επενδύσεις διότι από τη μία λέμε ότι το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων είναι ε, εν ζωή και λειτουργεί και από την άλλη τα αποτελέσματά του φοβάμαι λοιπόν ότι και η απουσία των συναδέλφων δεν οφείλεται στο ότι προηγήθηκε ένα καλό γεύμα αλλά γιατί δεν περιμένουμε και πολλά από αυτά τα οποία έχετε τουλάχιστον μέχρι τώρα κάνει. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, σύντομη η παρέμβασή Ήταν μεγάλη η παρέμβασή σας και θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομιλητές. Μάλλον να ακούσουμε τις απαντήσεις και ενδεχομένω και άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχά, ο κύριο Κόζα ε, ρώτησε για τι συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Είναι η πιο σημαντική υπηρεσία που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ήδη έχουμε λάβει 160 αιτήματα από υπευθύνου ε, project και τα πιο πολλά αιτήματα προέρχονται από τον ιδιωτικό κλάδο. Πάνε τα πράγματα μόνο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Για να δώσουμε λοιπόν υπηρεσίε στις δημόσιες αρχές, αλλά φαίνεται ότι ο ιδιωτικό κλάδος θέλησε να χρησιμοποιήσει τις ε, υπηρεσίες βουλευτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ από τις δημόσιες αρχέ. Άρα λοιπόν και ο δυτικό κλάδο ε, το βλέπει θετικά. Τα πιο πολλά αιτήματα δε συνδέονται με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου. Και πολλοί ρωτούν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, ε, ευρωπαϊκούς πόρους από τα ζωφεντικά ταμεία, τι σημαίνει η FSI και κατά πόσο μπορούν να συνδυαστούν οι πόροι. Κοιτώντα ε, το μέλλον τώρα των ε, συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνδυάσουμε την DigiRegia, DigiEcfin, DigiAP με καλύτερο τρόπο και να δώσουμε επιτόπου Τέτοιε υπηρεσίε συμβουλευτική. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είχαμε κάποιες ε, καλές ε, εμπειρίες. Η e IP και η DG ECFIN έχουν τονώσει την παρουσία τους στην Ελλάδα και για το λόγο λοιπόν αυτό η Ελλάδα κατάφερε να χρηματοδοτήσει με το EFSI τέσσερα ήδη έργα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι δημόσιες αρχές είναι μάλλον αργές σε ό,τι αφορά την κατανόηση του ΕΦΣΥ. Σε πολλές περιστάσεις, λοιπόν, τα μέλη του γραφείου μου έχουν ε, συναντηθεί με τις ελληνικές αρχές και έχουν δώσει συμβουλές και έχουμε πολύ καλές σχέσεις εργασίας με τις ελληνικές αρχές πλέον και πλέον πιο σημαντικό είναι αυτό ότι έχουμε καταφέρει να περάσουμε το μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πολύ βασικό αυτό. έχει παθιάσει το θέμα της ε, πλατφόρμας επενδύσεων στην ενέργεια, στον τουρισμό στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσε να συνενώσει πολλά μικρά project. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση ήταν πολύ βοηθητική σε ό,τι αφορά τη σύσταση τοπικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές, τις τοπικές αρχές. Αυτό προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να κοιτάμε δηλαδή τις βέλτιστες πρακτικές ανακατός μέλους. Το πρώτο έτος του ΕΦΣΗ Σας έδωσα ήδη κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αν θα θέλαμε να θέξουμε κάποια ζητήματα τα οποία μας απασχολήσαν και ποια είναι τα απορίσματα που, στα οποία καταλήξαμε σε ό,τι αφορά τις ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ειλικρινά σας ενθαρρύνω α, ως βουλευτές να κάνετε εκδηλώσεις και τέτοιες... Ε, να δίνετε ευκαιρίες ε, ενημέρωσης για το ΕΦΣΥ στις επικρατείες σας, γιατί πάντα στις περιπτώσεις αυτές το feedback είναι πάρα πολύ θετικό. είναι μεγάλο το ενδιαφέρον για το ΕΦΣΥ, για το επενδυτικό αυτό ταμείο. Αν οποιοδήποτε λοιπόν από εσά θα ήθελε και θα ενδιαφέρονταν να οργανώσει κάτι, Μπορεί να σας βοηθήσει η EIB, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που έχει γραφεία στα πιο πολλά, στις πιο πολλές χώρες και παρέχει βοήθεια στους βουλευτές, αλλά και η αντιπροσωπεία μας μπορεί να σας βοηθήσει με κάποια συνδρομή πληροφόρηση για τις εκδηλώσεις αυτές. Άρα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ακόμα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ε, μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτών και σε ορισμένε περιπτώσει μεταξύ και των δημόσιων αρχών για τη χρήση του ΕΦΣΑ. Του Ο κ. Πυρίνσκι έθιξε επαναλημμένα το θέμα της συνοχής στις κεντρικές ε, και ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαιτέρως, έχουμε ένα μεγάλο θέμα να εξηγούμε τι είναι το ΕΦΣΥ. Γιατί η πρώτη αντίδραση των δημοσίων αρχών είναι ότι δεν ενδιαφέρονται. Ενστικτοδός. Και έτσι δεν ακούν γρήγορα. Βάζουν παροπίδες και δεν μεταφέρουν το μήνυμα προς τον, δημο... προς τον ιδιωτικό κλάδο. και το ΕΦΣΙ κυρίως ε, στους ιδιωτικούς επενδυτές απευθύνεται. Εμείς έχουμε μάθει και εμείς το μάθημά μας. Έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένα με τέτοιες αρχές και λέμε για παράδειγμα, κοιτάξτε τι κάνουν οι γειτονικές χώρες, γιατί και εσείς δεν δραστηριοποιήσετε. Προσπαθούμε να δώσουμε καρά παράδειγματα σε ό,τι αφορά την συνδυασμό των πόρων και καλούμε τις κυβερνήσεις να είναι ενεργές για να βρουν, να εντοπίσουν καλά έργα και παρέχοντας τεχνική άρρωγη για την συντονισμό των πόρων. Οι χώρες ε, συνοχής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΕΦΣΥ εφόσον υπάρχει ομοσχετική επιθυμία. Τα έργα σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι χώρες ποιο ανετα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΕΦΣΥ μέσα στη χρηματοδότηση από τα δραστικά ταμεία. Και όπως είπα και εισαγωγικά, στη Βουλγαρία υπάρχουν ε, τρεις ειδικές τράπεζες που έχουν συμφωνήσει για την ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη Ρουμανία δεν υπάρχουν. Έχω δώσει και κάποιες συνεντεύξεις, έχω επισκεφθεί επανειλημμένως στην Ρουμανία και θα την ξανά επισκεφτώ για να εξηγήσω στους τραπεζίτες ότι για αυτούς είναι το εύση. Σε αυτούς απευθύνεται. Για να μην μακρηγορώ, χρειάζεται σε, διάφορες, σε διάφορα επίπεδα ε, ευαισθητοποίηση. Εξηγώντας τι κάνουν και οι άλλοι. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τι είδους ε, project έχουν χρηματοδοτηθεί με το ΕΦΣΥ, μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολύ ενδιαφέροντα πρόγραμματα που θα βοηθήσουν όλα τις μικρότερες επενδύσεις. Ο κύριος Πυρίνσκι έθεσε το θέμα της μεταρρύθμισης των επενδύσεων και των θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει σύνδεση όπως θα ξέρετε. Υπάρχει εξάντα αιρεσιμότητα στους ε, πόρους του ΕΦΣΥ, το οποίο και θα ενθαρρύνει τα κρατη να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Εδώ οι ανάγκες είναι διαφορετικές ανακρατός μέλος. Κοιτώντας όμως ε, τι χρειάζεται, για τι ε, θέσεις απασχόλησης ποιότητα ποιότητας μακροπρόθεσμα, μπορούμε να πούμε ότι σε, πολλά, σε πολλές χώρες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ε, κυρίως ό,τι αφορά τη βελτίωση τη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού συστήματο και της κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Εγώ αρχικά θεωρούσα ότι κάθε δάσκαλος, κάθε καθηγητής ε, στην Ευρώπη έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα, πτυχίο. Όχι όμως, από ό,τι φάνηκε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί μια απαραίτητη εκ των ουκάνευ προϋπόθεση για να υπάρχει καλή διδασκαλία, καλή εκπαίδευση. Και γι' αυτό είναι πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι επικεντρωνόμαστε σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και θα προωθήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Από τη βάση προς τα πάνω. Η συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και στο ΕΦΣΥ και γενικότερα στα επευετικά σχέδια. Προσπάθησα να εξηγήσω λίγο πολύ ποιες είναι οι προκλήσεις Δεν μπορούμε όμως να τα παρατήσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Για την συμπληρωματικότητα του ΕΦΣΥ, πολύ συχνά τίθενται σχετικά ερωτήματα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιλέγει τα προγράμματα, τα σχέδια. Ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί για κάθε σχέδιο που έχει εγκριθεί Ποιος είναι ο παράγοντας αυτός της συμπληρωματικότητας, προστατικότητας. Στις ε, πιο πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, είναι σαφέστατη αυτή η συμπληρωματικότητα. Είτε πρόκειται για σχέδια τα οποία δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν, είτε πρόκειται για σχέδια τα οποία δεν θα είχαν τις διαστάσεις και την ταχύτητα που σημείωσαν με το ΕΦΣΥ. Αλλά είναι πολύ βασικό αυτό. Πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων του ΕΦΣΥ. Είχατε και άλλα ερωτήματα τα οποία δυστυχώ δεν μπορώ να σα απαντήσω, αλλά θα τα θέσω στην Επιτροπο Κρέτσου για να σα τα απαντήσει γραπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έξι ερωτήσει έχουμε ακόμα και μετά πρέπει να ψηφίσουμε. Σε 35 λεπτά περίπου. Οπότε ελπίζω ότι θα είσαστε σύντομοι στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κυρία Αγγέα. Κοιτάξτε, αν ο καθένας μιλάει 10 λεπτά ένα τέταρτο, ε, τώρα οι υπόλοιποι που έχουν να μιλήσουν δεν θα έχουν το χρόνο για να θέσουν τα θέματά τους. Κύριε Επίτροπε, εσείς παρουσιάσατε ε, σε τέσσερα τμήματα αυτά τα οποία μας είπατε και αυτό προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Καταρχάς, οι ικανότητες, ε, <clears throat> λέτε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων και ανάγκη διαφθρωτικών αλλαγών. Μιλήσατε επίσης ε, για την επαγγελματική κατάρτιση, για τα για τα στάζ επίσης, τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, αλλά δημιουργούν προβλήματα, γιατί στην ουσία εκμεταλλεύονται τους νέους σαν εργαζόμενους χαμηλού κόστους και όχι σαν ένα πραγματικό μέσο απόκτησης γνώσεων. Τώρα για την κατάρτιση αυτών που με τη σειρά τους καλούνται να καταρτήσουν τους υπόλοιπους. Και εδώ στις προτάσεις αναχώρα ζητάτε ε, αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση, όμως τα τελευταία μέτρα έχουν καταστραφεί θα έλεγα τα σχολεία δυστυχώς είχαμε εξαιρετικά συστήματα και είπατε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε άλλα συστήματα εκπαιδευτικά, ενώ θα έπρεπε τα άλλα να ταυτιστούν με τα δικά μας. Γιατί ήταν διεθνώς αναγνωρισμένα τα συστήματά μας στην επαγγελματική κατάρτιση, ήταν κατάλληλα όχι μόνο για την προετοιμασία των σπουδαστών, αλλά και για τη δημιουργία προϋποθέσεων για σωστή εργασία αυτών που διδάσκουν. Οι δυνατότητες χρήσης των μεταναστών θα συμφωνήσετε με την στάση σαν παράδειγμα της Γερμανίας η οποία προσφέρει 2 ευρώ την ώρα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας οι μετανάστες. Εγώ αυτό το ονομάζω εκμετάλλευση και δεν είναι κάτι το οποίο ε, λύνει το πρόβλημα της απασχόλησης για το στρατηγικό ε, ταμείο. Ε, είπατε να κοιτάξουμε τα tweet τα οποία κάνετε σε ποσοτικό επίπεδο. Ε, για την Ιταλία υποθέτω ότι μπορεί να είναι θετικά, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν οκτώ προγράμματα, το ένα πιο επικίνδυνο από τα άλλα, πολύ ρηψοκίνδυνα και οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές που θα πάρουν χρήματα λειτουργούν με πελατειακό τρόπο, κάτι το οποίο πρέπει να σας κάνει να είσαστε πιο προσεκτικοί και επακριβείς. Και τέλος για το χάλιβα. Εγώ είμαι από την Όμπρια, Ξέρετε την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, Thyssen Group, το εργοστάσιο αυτό, το χαλιβουργείο το οποίο υπήρχε, που ενέπλεξε και την ιστορία για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Έχουμε ένα σύστημα εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη στρεβλό, γιατί δεν έχουμε αποτελεσματικές βιομηχανικές πολιτικές με οράματα για το μέλλον. <clears throat> Από την άλλη, εμείς στην Ιταλία έχουμε δει, μείνει με δύο μόνο μεγάλες εταιρείες και διαρωτώ με αν δώσουμε την ε, ιδιότητα της οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, τότε τι θα γίνει με τη βιομηχανία μας, η οποία ήταν εξαιρετικός παραγωγός, ήμασταν αναγνωρισμένοι παγκόσμια και η δική μου χώρα είχε ένα συγκεκριμένο πλούτο, δυστυχώς όμως τον καταστρέψαμε τον πλούτο αυτό, δυστυχώς και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων στα εργοστάσια αυτά οι συνέπειες ήταν πολύ κακές από τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τα λάθη γιατί δεν έχουμε ένα όραμα βιομηχανικής πολιτικής. Εσείς είπατε ότι είστε διατεθειμένος να μιλήσετε για το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων στα κράτη-μέλη. Εγώ θέλω να σας προσκαλέσω στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Όταν μιλάμε για μεγάλες υποδομές σε μια χώρα σαν τη δική μου, από τις πιο πλούσιες και όμορφες στον κόσμο, στην ουσία καταστρέφουμε αυτά που έχουμε. Και θα πρέπει να έρθετε μαζί μας για να δώσουμε εξηγήσει ε, ε, στους πολίτες ότι δυστυχώς δεν δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης, δυστυχώς δεν δημιουργείται από τις μεγάλες επενδύσεις απασχόληση, είναι στιγμιαία αν τυχόν δημιουργηθεί, όταν σταματήσει να λειτουργεί δηλαδή πάβει και η δημιουργία των θέσεων και νομίζω ότι απαιτείται να έχουμε ένα συνολικό όραμα για το τι θέλουμε Είχαμε ένα όραμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετατρέψαμε τις πολεμικές βιομηχανίες, δημιουργήσαμε τέρατα βιομηχανικά βέβαια, κάποια από αυτά που ακόμα και σήμερα σκοτώνουν τους ανθρώπους που κατοικούν γύρω και δεν δημιουργούνται ταυτόχρονα σημαντικοί αριθμοί θέσεων απασχόλησης. Ο, ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Ήρθατε να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητές σας και σας ευχαριστούμε. Μεταξύ άλλων αναφερθήκατε στη Χαλιβουργία ως προτεραιότητα. Μέσω λοιπόν αυτού του στρατηγικής σημασίας κλάδου, γιατί όχι μόνο έχουμε χάλιβα, αλλά γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα της απασχόλησης, των αμοιβών, το θέμα της έρευνας, της καινοτομίας και οι επενδύσει είναι αυτά που μα ενδιαφέρουν. Και τα λέω αυτά γιατί όταν εσεί λέτε ότι έχετε ένα σύστημα ελέγχου των εισαγωγών χάλιβα, κυρίω των κινέζικων, αν έχετε τέτοιο σύστημα ελέγχου είναι μάλλον κακό, γιατί 2 εκατομμύρια τόνοι έρχονται. Το 2015 είχαμε 37 εκατομμύρια τόνους κινέζικου χάλιβα που μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και για πρώτη φορά στην ιστορία μας, για πρώτη φορά, η Ευρώπη ήταν ελληματική σε σχέση με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και πράγματι αναφερθήκατε στο πρόβλημα της τιμής του, γιατί το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε ζήτηση, το πρόβλημα είναι η τιμή. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας, ε, ούτε μία βιομηχανία στον κόσμο, ούτε καν η Κίνα που κερδίζει από το χάλιβα. Χάνουν οι Κινέζοι 55 δολάρια ανά τόνο ε, χάλιβα που παράγουν. Και στην Ευρώπη πουλάμε στην τιμή της πρώτης ύλη. Πού είναι λοιπόν το κινέζικο θαύμα. Η συνεδρίαση του ωσά εγώ ήμουνα σε αυτή την συνάντηση και οι Κινέζοι δεν ήρθαν για να κάνουν διάλογο ή διαπραγματεύσεις μαζί μας, ήρθαν για να μας εκφοβήσουν, ήρθαν για να μας πούμε πρόσοχη τι θα κάνετε. Και ήσασταν στην Κίνα και η κυρία Μέρκελ πήγε πριν από, δε, από κάμια δεκαριά μέρες για να θέσει το θέμα αυτό της υπερβολική παραγωγής χάλιβα από την Κίνα. Όταν λοιπόν έφτασε στην Κίνα, πολλά χαλιβουργία ξανάρχισαν στην Κίνα. Οπότε η δέσμευση της Κίνα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσει την παραγωγή τη δεν είναι αλήθεια. Οπότε πώς θέλετε να έχουμε και το επίπεδο ε, θέσεων απασχόλησης ε, ποιότητας. Όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, έπειτα για την καινοτομία, το ίδιο. Υπάρχουν ε, χίλιες παραλλαγές στην, στον κόσμο που δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι η καινοτομία λοιπόν είναι τεράστια στον κλάδο. Όμως με αυτό το ρυθμό σε λίγους μήνες δυστυχώς μπορεί να εξαφανιστούμε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε τον κινέζικο ανταγωνισμό. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τις προσπάθειες, όχι απλώς να ελέγχουμε τις κινέζικες εισαγωγές, αλλά επίγει να έχουμε μέτρα αντι-dumping, όπως κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν 300% ε, σχεδόν ε, φόρο, για να μην έχουν ζημιά. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο πριν που αναφέρθηκε και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα αυτά που προετοιμάζουμε δεν προστατεύουν αρκετά. Πρέπει να προστατεύσουν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τους εργαζόμενους. Αν όμως το μόνο που θα κάνουμε είναι να επιβάλλουμε παραπάνω φόρους στου, στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, θα εξαφανίσουμε πιο γρήγορα ακόμα ένα κλάδο που είναι ζωτική σημασία για την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομος αυτή τη φορά από ό,τι ήμουν πριν. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο θέμα των νέων που λέτε ότι γίνεται κατάχρηση, ότι τους χρησιμοποιούμε για φτηνό εργατικό δυναμικό, αντί να χρησιμοποιούμε άλλους με πολύ υψηλότερα προσόντα και καταρτισμένους καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομοθεσία. Είναι εθνική αρμοδιότητα. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν τους ε, εργασιακούς τους νόμους και το τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό και που είναι το όριο ανάμεσα στο internship, την ε, μαθητεία, τα στάζ και ένα, μια πραγματική σύμβαση εργασίας. Συνεπώς είναι δύσκολο για μας να πούμε οτιδήποτε στις χώρες μέλη από αυτού. Γενικότερα όμως, δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνει κανείς τη διάκριση ανάμεσα σε μια μόνιμη εργασία ή μια κανονική σύμβαση εργασίας και την μαθητεία. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις χώρες μέλη να χρησιμοποιούν την μαθητεία όταν έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ανεργία. Αυτός ο τρόπος μαθητής είναι πολύ καλός για να εισαχθεί κανείς και στην αγορά εργασίας και για να κάνει κάτι, για να μην μείνει χωρίς τίποτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιείται, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι το καθεστώς αυτό δεν πρέπει να στρεβλώνει την βιώσιμη αγορά εργασία. Η Ευρώπη έχει πολλές καλές πρακτικές από αυτού και στις χώρες που θεωρεί κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να κοιτάμε τις βέλτιστες πρακτικές στις άλλες χώρες. Για τη Χαλιβουργία. Το θέσανε πολύ. Θα συνδυάσω λοιπόν τις δύο ερωτήσεις. Η Κίνα έχει ικανότητα παραγωγής χάλιβα μεγαλύτερη από ό,τι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό πάντα dumping. Όμως, προφανώς, αν υπάρχει τόσο μεγάλη ικανότητα παραγωγής, κάπου πρέπει να το πουλήσεις. Και άρα πρέπει κάτι να κάνεις με την τιμή. Και εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος του dumping. Δεν έχω τα ακριβή στοιχεία στο μυαλό μου, έχω όμως κάποια νούμερα υπόψη μου για το μερίδιο του κινέζικου χάλιβα που υποβάλλεται στα μέτρα αντιντάπινγκ. 17% του κινέζικου χάλιβα είναι κάτω από αυτά τα μέτρα κατά των ε, επιδοτήσεων. Δεν έχω βέβαια την ακριβή απάντηση στο μυαλό μου, αλλά όταν λέτε ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξέρετε ότι τα χρησιμοποιεί κάθε φορά όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θέτουν το ζήτημα και αναλύουμε τις διάφορες περιπτώσεις, οπότε αποφασίζουμε την ε, ξένη επιχείρηση, να τη θέσουμε, να μην τη θέσουμε υπό τα μέτρα αυτά. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν πιο γρήγορα από ότι εμείς. Αλλά θα αλλάξουν και τα δικά μας αμυντικά εμπορικά μέτρα και θα μπορούμε πιο γρήγορα να τα χρησιμοποιούμε. Υπήρχε επιχείρημα από τις χώρες ε, μέλη Βέβαια υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν λέω ότι όλα έχουν προχωρήσει. Κάποιες χώρες αντιδρούν ακόμα. Από εκεί και πέρα το Συμβούλιο θα αποφασίσει τι είναι διαφορετικό ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη όσον αφορά το αντιτάπινγκ και μέτρα κατά των επιχορηγήσεων είναι ότι πιο συχνά αποφασίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε από την Ευρώπη. Και πιο συχνά πάνε στο δικαστήριο από την Ευρώπη. Βελτιώνουμε πάντως το σύστημά μας και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το δίκαιο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και τηρεί κάποιες αξίες όσον αφορά το εμπόριο. Θέλει πιο ανοιχτό εμπόριο, πιο δίκαιο εμπόριο. Αν θέλετε να είσαστε πιο ανοιχτό στο εμπόριο, συγχρόνως πρέπει να είσαστε διατεθειμένος και να εφαρμόσετε δίκαια εμπορική πολιτική. Το ελεύθερο εμπόριο δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Μερικές φορές ζημιώνεστε και γι' αυτό πρέπει να είσαστε πάντα σε θέση να υποστηρίξετε και τα δικά σας συμφέροντα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ντομινίκ Μαρτά και συγγνώμη που μπερδεύτηκα προηγουμένω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την παρέμβαση της Λάουρα ήθελα να πω ζήτω η Ιταλία και μετά από την παρέμβαση του Εντουάρ Μαρτά να του πω ότι υπάρχει κι άλλος Μαρτάν σε αυτή την αίθουσα και ότι τώρα τον λόγο τον έχει ο Ντομινίκ. Αλλά αγαπητέ Εντουάρ, ενθουσιάστηκα, ενθουσιάστηκα γιατί έμαθα ότι επιτέλους είστε υπέρ ε, μιας λογικής μορφής προστατευτισμού. Ιδιαίτερα όταν φύγονται τα συμφέροντά σας. Στο παρελθόν δεν το κάνατε αυτό τώρα ξαφνικά ο χάλιβας σας ε, ενδιαφέρει και θέλετε να υπάρξει προστατευτισμός για το χάλιβα και τόσο το καλύτερο. Τώρα κύριε Αντιπρόεδρε Κατάιναν πρέπει να ομολογήσω ότι ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο κάνατε την παρέμβασή σας κόντεψε να με ξυπνήσει. Να σας πω βέβαια ότι εσείς έχετε ουσιαστικά την εξουσία εδώ και δεκαετίες. Η Επιτροπή είναι, αν θέλετε, η ηγέτης εισαγωγικά για τα θέματα αυτά εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά για τα οποία παραπονιέστε, έλλειψη ικανοτήτων, αναλφάβητη, 25% των ενηλίκων χωρίς δίπλωμα, ε, είστε και υπεύθυνοι γι' αυτά. ακόμα και στα πλαίσια του διαρθρωτικού διαλόγου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2016. Στην ουσία αγνοείτε το τι κάνατε τα τελευταία 30 χρόνια. Μας μιλάτε για το πρόγραμμα επενδύσεων λέγοντας ότι θα αναχρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες. Ε, τις τράπεζες, εντάξει. Οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, και οι ιδιώτες δεν θέλουν οι τράπεζες να αναχρηματοδοτηθούν. Θέλουν οι ίδιοι να αναχρηματοδοτούνται γιατί αυτοί έχουν ανάγκες. Οι τράπεζες δανείζουν χρήματα και είναι κρίμα αυτό που κάνετε. Τώρα για το χάλιβα μιλήσαμε επί μακρόν, δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο. Και τώρα σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα κύριε Αντιπρόεδρε, το να ξεκινάτε διαβουλεύσεις είναι φρούδες ελπίδες και λέτε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά ταμεία και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να ανακουφίζουν τους εργαζομένους. Από τη μία λοιπόν κάνετε ό,τι μπορείτε για να εξαφανίζονται οι επιχειρήσεις μας ή να το πω αλλιώ, δεν κάνετε τίποτα για να μην εξαφανίζονται. Και από την άλλη ο κόσμος εξεγείρεται και εσείς αυτό το ονομάζετε λαϊκισμό και στέλνετε εκατομμύρια στις διάφορες επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 500 εργαζομένους. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή η πολιτική σας. Ο κύριος Μπερνίτσκι είχε και αυτός, ε, ο κύριος Πυρίνσκι εννοεί μάλλον ο κύριος Μαρτά, ε, παρότι ανήκει σε μία από τις μεγάλες ομάδες ε, στο Κοινοβούλιο που υπαγορεύει τις πολιτικές εδώ και 30-40 χρόνια, στην ουσία αυτό το οποίο έκανε ήταν να επιτεθεί εναντίον σας και να, θα έλεγα, να οδηγήσει σε κατάρρευση το πρόγραμμά σας. Ε, εντάξει, εσείς μας είπατε τώρα παρακολουθήστε τα tweet για τα ποσοτικά στοιχεία. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, tweet. Τώρα αυτό το πιστεύετε. 21 Ιουνίου του 2016. Ε, τώρα αυτό είναι λίγο φτωχό. Λοιπόν, φανταστείτε το σύνολο των πολιτών στην Ευρώπη να ακούσουν αυτό το οποίο είπατε. Ακολουθήστε με ε, στα Twitter. Ε, τώρα σωθήκαμε. Λοιπόν, ο κύριος Πυρίνσκι, λέει ο κύριος Μαρτά, αλλάζοντας πάλι το όνομα, ε, πράγματι υπήρχε κάτι το δυναμικό στην παρέμβασή σας. Θα τελειώσω γιατί έχω μιλήσει σχεδόν πέντε λεπτά για το κοινωνικό ντάμπινγκ κουβέντα. Ε, για το TTIP, ενώ είναι στο πρόγραμμά σας ε, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, Ισορροπή και ε, έλογη με τις Ηνωμένε Πολιτείες και συνεχίζεται τις διαπραγματεύσεις. Ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεχθείτε το TTIP τελειώσαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε ένας έξυπνος νέος κύριε ε, Αντιπρόεδρε, αλλιώς δεν θα ήσασταν εκεί που είσαστε. Η ερώτησή μου είναι απλή. Μήπως τελικά αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας το τιμόνι του Τιτανικού κύριε Αντιπρόεδρε. You have finished. Ολοκληρώσατε λοιπόν και θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ριμπέρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να είμαστε ευγενείς προς τους προσκεκλημένους μας, ε, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε προσβολές προς έναν επίτροπο, προς έναν προσκεκλημένο, ο οποίος έχει έλθει να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις. Προσβάλλοντας τον επισκέπτη μας, δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Μα σε ποια φάση ε, προσέβαλα και φτάνει πια με ε, ε, τα διδάγματά σας. Ήμουν ορθώς και είπα ότι αν δεν υπάρχει, σταματήστε λέει η Πρόεδρος. Κανείς δεν είναι παρόν και δεν ξέρουμε γιατί. Αν θέλετε λοιπόν τα μαθήματά σας και τα διδάγματά σας να κρατήσετε για τον εαυτό σας κύριε Κάζα και διακοπτή πρόεδρος ε, κυρία Ριμπέιρο, ε, πάρτε το λόγο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες αυτή τη στιγμή μαζεμένοι εδώ στην αίθουσα. Μα ναι, όχι, θα με, θα με κρίνει εμένα ο κύριος Κάζα. Η κυρία Ριμπέιρο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, λέει κυρία Ριμπέιρο, είναι... Α, θέλει να πάρει το λόγο κύριο Μαρτά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας πω το εξής κυρία Πρόεδρε. Ως ε, δασκάλα και ως μέλος συνδικάτου ήμουν πολύ ικανοποιημένη με τις προτεραιότητες που θέσατε. Καταρχάς, ε, με την ανάγκη να δημιουργηθούν πιο πολλές συγκεκριμένες δεξιότητες στο πλαίσιο της ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρέπει να ομολογήσω, Αντιπρόεδρε, ότι δείξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να αναγνωρίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα επιλύσουμε βράχη πρόθεσμα. Γιατί ο αντίκτυπος θα φανεί μέσω και μακροπρόθεσμα. Ιδάλλως ε, θα δούμε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία, λίγο τυχαία αν θέλετε, από πλευρά των κρατών μελών, τα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν την εντύπωση ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σε ό,τι αφορά τα καλύτερα αποτελέσματα με την εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να θέσω εδώ, σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, το ότι είναι σημαντικό το ότι τονίσατε το θέμα της εκπαίδευσης των δασκάλων και καθηγητών. Αυτό δεν μπορεί να έχει να κάνει ασφαλώς μόνο με, τις πρώτες, με τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης. Όχι, θα πρέπει να ισχύει και στην διαβίου μάθηση σε όλες τις καριέρες ε, σε βάθος 30-40 ετών. Θα πρέπει λοιπόν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να ενημερώνονται, να επικαιροποιούν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους. Αυτό σημαίνει φυσικά με τη σειρά του επενδύσεις. Άρα, θα πρέπει να αντιστρέψουμε κάποιες από τις προτεραιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης των δασκάλων. Κάποιες από τις προτεραιότητες οι οποίες προωθήθηκαν από τα πρόσφατα χρόνια. Τελευταία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των κρατών μελών στο ΕΦΣΥ, σας ερωτώ, πώς ε, θα δημορφωθεί αυτή η αερογενική συνεισφορά. Πολύ σημαντική λοιπόν η πρόσβαση στο ΕΦΣΙ και γι' αυτό λοιπόν η σχετική έκκληση ε, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιμετωπίζω μεγάλε δυσκολίε σε ό,τι αφορά και τι απόκεντρε ε, περιοχέ. Κύριε Επιτροπέ, θα μπορούσατε να μα βοηθήσετε. Θα εκτιμούσα Ιδιαίτερα θα σε, ήθελα να σας καλωσορίσουμε και στις Αζόρες ε, για να συναντηθείτε και με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εκπροσώπους του κόσμου, ε, να δώσετε πληροφορίες προκειμένου να συμμετέχουμε και εμείς στο σχέδιο αυτό. Και μία νότα αισιοδοξία είμαι εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για την έκθεση που συζητήθηκε το Φεβρουάριο και για την γνωμοδότηση που θα παρουσιαστεί αύριο. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω με θετικό πρόσημο το γεγονός ότι τονίζεται ο κοινωνικός διάλογος, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Τίθεται θέμα βιωσιμότητας του κρατούς, των εθνικών κρατών και την βιωσιμότητα των, ε, της ε, το ευρωπαϊκό μοντέλο, Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, λοιπόν, όπως ε, το γνωρίζουμε, ενδεχομένως να διακυβευτεί στο μέλλον. 7%, 7 του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να μετρηθεί, λοιπόν το μοντέλο αυτό και θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλα όσα έχετε κάνει προς την κατεύθυνση αυτή της ε, συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάντερ. Συγγνώμη. Ο κύριος Εμίλιαν Πάβελ. Είναι περίπλοκος ο κατάλογος ε, σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Αντιπρόεδρο που βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί ήδη αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα τα οποία ήθελα να σα ε, θέσω. Να είμαστε λίγο πιο ακριβείς για την κατάσταση στην Ρουμανία. Είπατε και δίκιο έχετε ότι δεν είναι οι τράπεζε που παρέχουν τέτοια προγράμματα επενδύσεων. Είπατε επίση ότι θα έχετε πιο πολλές επικοινωνίες με τις τράπεζες για να συμπεριληφθούν στα προγράμματα αυτά. Θα σας σύστηνα να συζητάτε πάντα με τις μητρικές τράπεζες. Τράπεζες ε, στην Αυστρία, στην Γερμανία, στη Γαλλία, γιατί στην Ρουμανία έχουμε μόνο μία αμυγός ρουμανική τράπεζα. Ξέρω ότι διοργανώθηκε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μας τον Φεβρουάριο πρώην Επίτροπο, άλλωστε, θα πρέπει να καταλαβαίνει τη σημασία των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα μπορούσατε να μας ε, ενημερώσετε για το τι συζητήσατε και ποια είναι τα προβλήματα, γιατί η Ρουμανία δεν λειτουργεί σωστά σε αυτό το επισημαντικό πρόγραμμα. Τέλος. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να διοργανώσετε πιο πολλές εκδηλώσεις στην ε, Ρουμανία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ε, νέους εκλεκθέντες ε, δημάρχους ε, που θα εφαρμόσουν τα προγράμματά τους για την επόμενη τετραετία. Σας ενθαρρύνω λοιπόν και θα χαρώ να σας βοηθήσω αν χρειαστεί η την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα η κυρία Σαντέρ. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ σήμερα και εγώ σε αντίθεση με κάποιους συναδέρφους ή κάποιον ο οποίος δεν είναι πια εδώ έφυγε, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αλλάξει ε, τα πράγματα μαζί με εμάς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να βελτιωθεί η απασχόληση στις διάφορες χώρες μέλη. Αναφερθήκατε σε διάφορα σημεία. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να επιμείνω στις ε, ικανότητες, τις ε, δεξιοτεχνίες τις οποίες αναφερθήκατε. Από τη μια έχουμε την απόκτηση των ικανότητων αυτών και εδώ συμφωνώ με τις διάφορες λύσεις που προτείνεται ότι πρέπει να παρεύουμε σε επίπεδο εθνικής εκπαίδευσης πρώτα απ' όλα. Θέλω Επίση να τονίσω και το θέμα της στήριξη της κατάρτιση, γιατί μπορούν με τέτοια κατάρτιση επιχειρήσεις οι νέοι μας να έχουν το ένα πόδι στην εκπαίδευση και το άλλο ε, στι επιχειρήσει. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Πρέπει επίση να αναπτυχθεί περισσότερο και το πνεύμα ε, του επιχειρήν, γιατί είναι και αυτή μια γνώση, μια ικανότητα που μπορεί να βοηθήσει τους νέους να φτιάξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Ή όχι, αλλά αν μη τι άλλο θα ξέρουν πώς να το κάνουν, αν θέλουν να το κάνουν. Πέρα λοιπόν από την απόκτηση των ικανοτήτων υπάρχει και το θέμα της αναγνώρισης όμως των προσόντων, των γνώσεων. Εγώ έρχομαι από μια διασυνοριακή περιοχή από την Αλσατία. Έχουμε δίπλα μας τη Γερμανία. Στην Αλσατία έχουμε υψηλή ανεργία. Από την άλλη μεριά των ε, συνόρων υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Γίνεται λοιπόν πολλή δουλειά επιτόπου ώστε να προσφερθεί η κατάλληλη κατάρτιση στους νέους Γάλλους, ώστε να μπορούν αυτοί να βρουν δουλειά στη Γερμανία στη συνέχεια. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αναγνώριση των προσόντων τους, γιατί οι Γερμανοί επιχειρηματίες δεν κατανοούν τι προσόντα διαθέτουν αυτοί οι νέοι που έχουν γαλλικά διπλώματα. Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, ρωτάω, τι μέσα έχουμε για να προχωρήσουμε στο θέμα της αναγνώρισης προσόντων και διπλωμάτων αμοιβαία. Απάντηση, παρακαλούμε κύριε Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Μαρτά. Έφυγε. Αν ήταν εδώ, θα το έλεγα. Ντομινίκ Μαρτάν, γιατί έχουμε δύο Μαρτάν στην αίθουσα, να μην μας μπερδεύετε παρακαλώ. Έτσι, γιατί και εγώ είμαι Μαρτάν, μην με μπερδεύετε με τον άλλο Μαρτάν. Και εγώ είμαι στην αίθουσα. Κατά είναι. Ναι, είναι εύκολο να ακούει κανεί την κριτική ότι όλα έχουν γίνει στραβά και όταν ήταν το κόμμα του και στην εθνική κυβέρνηση και στην Ευρώπη θα ήταν καλύτερα. Κοιτάξτε, κάποιε από τι επικρίσει δικαιολογούνται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πιο ειλικρινές αν εξηγούσε και αυτό στον κόσμο ποιες είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιες είναι αρμοδιότητες των χωρών μελών. Αλλά βέβαια θα του χάλαγε την ιστορία κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο. Το ΕΦΣΙ, το επενδυτικό ταμείο, δεν χρηματοδοτεί τράπεζες. Είναι αντίθετο προς την ε, ρύθμιση δημιουργίας του. Οι τράπεζες είναι αυτές που χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλιώς καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχαν εκατομμύρια αιτήσει και θα ήταν κακό για τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν έπρεπε να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όχι, είναι οι εθνικές τράπεζες που επενδύουν τις, που χρηματοδοτούν μάλλον τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορώ να σας δώσω. Κύριε Ριμπέιρο, η εκπαίδευση είναι μια μακροχρόνια επένδυση πράγματι. Αν δείτε την ψηφιοποίηση, ήδη βλέπουμε πώς έχει αλλάξει το τοπίο και ποιες είναι οι προκλήσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε αυτήν την μεταβιομηχανική εποχή. Εννοείται ότι μία λύση δεν είναι καλή για όλους. Αλλά οι χώρες μπορούν να μάθουν η μία από την άλλη. Το ΕΦΣΙ τώρα και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το μέγεθος της αγοράς. Καμιά φορά είναι δύσκολο να βρουν χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ΕΦΣΙ δίνει περισσότερες δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πιο απομακρυσμένων περιοχών χρειάζεται συνειδητοποίηση των τραπεζών που είναι παρούσες στις απομακρυσμένες περιοχές και γι' αυτό τους λέμε κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει το ΕΦΣΥ γιατί τότε μπορούν να έρθουν σε επαφή με το πιο κοντινό γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να ζητήσουν βοήθεια. Έπειτα, χωρίς βέβαια να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις αζόρες, πρέπει να σας πω ότι μπορεί να υπάρχει μια επενδυτική πλατφόρμα όπου το εύση να δώσει κάποια ποσά και να υπάρξουν κάποια επενδυτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις χώρες μέλη Σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει για ενεργειακά προγράμματα. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα μπορούσαν για τον τουρισμό να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια μέθοδο. Ναι, θα έρθω σε επαφή με τράπεζες στη Ρουμανία όταν μου δοθεί η ευκαιρία πάλι. Ναι, στην ε, Βουλγαρία έχει γίνει, δεν θυμάμαι τώρα με ποια, αλλά συμβαίνει. Έχουμε επίσης συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών που αντιλαμβάνονται απόλυτα το νόημα του επενδυτικού ταμείου και τους έχουμε ενθαρρύνει να κοιτάξουν και προγράμματα άδρευσης και να μπορούν άρα να χρησιμοποιήσουν το νερό το οποίο μπορούν να συλλέξουν όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις. Έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει ένα καλό πρόγραμμα άρδρευσης. Και η χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χρήματα από το ΕΦΣΥ. Και έτσι να εξοικονομήσει χρήματα από άλλες επενδύσεις για άλλους σκοπούς. Κυρία Σάντερ, η αναγνώριση των προσόντων, των ικανοτήτων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ενιαίας αγοράς. Αν θέλει κανείς να έχει μια ενιαία εργασιακή αγορά, αυτό πρέπει να το κάνει. Και το παράδειγμα που μας δίνετε εσείς είναι πολύ καλό. Ακόμα και εκεί που υπάρχει η συνήθεια νοοτροπία αυτή να πηγαίνει ο κόσμος και να δουλεύει στην γείτονα χώρα, παρόλα αυτά η αναγνώριση δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Η Επιτροπή λοιπόν πιέζει για την αναγνώριση, αλλά βέβαια όλα εξαρτώνται από το πώς υλοποιούν ε, τέτοιου είδους ε, ιδέες οι εθνικές αρχές. Μεταξύ Φιλανδίας και Σουηδίας, για παράδειγμα, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι τοπικές αρχές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο. Ακόμη και αν αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από τους υπουργούς, αλλά οι τοπικές αρχές αρχίζουν και συγκρίνουν πόσο διαφέρουν τα σχολικά προγράμματα μεταξύ των δύο χωρών. Και μάλιστα έβαλαν και τους επιχειρηματίες να καθίσουν ε, στο τραπέζι για συζήτηση και τους έβαλαν να πούνε τι προσόντα να ζητούν εκείνοι για να προσλάβουν ε, προσωπικό, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα το σχολικό πρόγραμμα κάθε φορά. Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν, ακόμα και σε πιο χαμηλό επίπεδο, όχι πάντα στο εθνικό. Είναι ένα καλό κακό παράδειγμα θα έλεγα, ότι και στην Αλυσατία υπάρχει αυτό το πρόβλημα της αναγνώρισης σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τα σχόλιά σας και ας συνεχίσουμε αυτή την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε λέει πρόεδρος. Are you ready to vote? Είμαστε έτοιμοι για τις ψηφοφορίες, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω στον κύριο Λαβριγιό και στον κύριο Κάζα ότι κάπου κάπου πρέπει να πηγαίνω στην τουαλέτα ε, πριν τις ψηφοφορίες. Oui, ε, γενικά έχει κάποια θέματα φαίνεται φυσιολογικού τύπου ε, και μπορεί να βγαίνει όποτε θέλει και να κάνει αυτό το οποίο θέλει κάθε φορά. Αλλά όταν είμαστε βουλευτές και μιλάμε τόσο άσχημα για κάποιους ανθρώπους, ε, ας μείνουμε για την απάντηση. Ε, λυπάμαι που δεν μπόρεσε να αναβάλει για λίγα λεπτά την τόσο σημαντική του αποστολή που τον οδήγησε εκτός εθούσης. Αλλά νομίζω ότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται με πολύ δημοκρατικό τρόπο. Και σύν της άλλης μας ζάλισε για πολλή ώρα για το ότι νίσταζε και ότι κανένας δεν τον ξύπναγε. Νομίζω ότι ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, και πολλές φορές ε, όταν ιστάζει κανείς μετά το μεσημέρι, μετά το φαγητό, ίσως να οφείλεται στο ότι έφαγε επί μακρόν, να το πω έτσι, και θα μπορούσε αν έτρωγε λιγότερο να κάτσει να ακούσει τον Επίτροπο ο οποίος ε, ε, είπε αυτά που είπε. Ε, λόγω του παρελθόντος του πολιτικού του κυρίου Λαβριγιώ εγώ χαίρομαι που πήρα μαθήματα, εμένα ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί μου η δικαιοσύνη. Τώρα, ε, Τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες, λέει η Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Τελείωσε αυτή η συζήτηση. Η κυρία Τζεπαλοβά έχει μία ερώτηση να κάνει για ένα άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ. Δεν θα συζητήσω φυσιολογικά και σωματικά θέματα, αλλά διαδικαστικά. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την διαδικασία που ακολουθείται και έγινε καταρτιστή η ερώτηση την οποία θα ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στην αρχή τη εβδομάδα ορίστηκαν οι υπεύθυνοι για την ερώτηση για την ε, πρωτοβουλία για την νεολαία. Είχε συμφωνηθεί για το περιεχόμενο ε, του, της ερώτησης με mail. Και προτείναμε λοιπόν το κείμενο αυτό στους συναδέλφους για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε στην τελική ψηφοφορία. 8, 8 το βράδυ ο κύριος Χάντελ άναξε μόνο μερός ε, το κείμενο της ερώτησης χωρίς διαβούλευση καμία με τους κοιόδες. Και τώρα, λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ψηφίζουμε το θέμα αυτό. Δεν θέλω κάποια απάντηση και ξέρω ότι θα υποστηρίξω την προφορική ερώτηση, αλλά πραγματικά να πιέμαι για τη διαδικασία από που ακολουθήθηκε. Η προφορική ερώτηση, δηλαδή, πλέον τι, καταρτίζονται μόνο από την Πρόεδρο και δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν οι σκιώδεις. Αυτό λέμε. Ε, Σας ευχαριστώ. Εξ όσων κατάλαβα υπήρξαν κάποια θέματα για το ζήτημα αυτό. Όπως και να έχει θα ψηφίσουμε τώρα. Γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Πρέπει να υποβληθεί το ερώτημα στον, ε, στην του Ιουλίου. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση. Πέρας. 42 υπέρ. Καμία αποχή. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε δικά ψηφοφορία για εσάς όμως, καταλαβαίνετε. Επόμενο ζήτημα, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Επόμενο θέμα σχέδιο σύσταση από την κυρία Γασλοβιέσκα για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ελβετίας σε ό,τι αφορά την προσχώρηση της Κροατίας. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου σύστασης ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Έχουμε μία ψήφο υπεράριθμη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. 45 υπέρ, 2 κατά. Τελική ψηφοφορία, επίσης ηλεκτρονικά. Πέρας. 44 υπέρ, 2 κατά. Να πάμε στην ε, οδηγία για την ισότητα της απασχόλησης τώρα. 56. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1β. Η 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Έλεγχος. Έλεγχο θέλετε. Για την παράγραφο 1β λίμπε 4. Ψηφίζουμε. Ψηφίζει ένας παραπάνω από το έλικο. Έναρξη. Και πέρας ψηφοφορίας. Πάλι περισσεύει ένας. Περισσεύει ακόμα ένας. great. Ωραία. Πέρασε. Εγκρίνεται 31 ψήφι υπέρ. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έναρξη. Συμβαστική 10. Oh, sorry. Sorry. Amendment. Συγγνώμη την 58, 59 και 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. open and now it is closed. Έναρξη και πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβαση και 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά Αποχές. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι υπερισχύουν οι αποχές. Για την 79 παρακαλώ, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Μία ψήφος παραπάνω από το ΕΛΚ. Είκοσι υπέρ. Εγκρίνεται. 14 είναι οι εποχές. Πάμε τώρα στην σεμιβαστική 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά Άποχες. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 ναι, 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7α. Η τροπολογία υπερθμών 100 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 101 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 103 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 25 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά Χρειάζεται έλεγχος για την 130. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Από το ΕΛΚ πάλι περισσεύει ένας. Τώρα είμαστε εντάξει. Οριακό. Το αποτέλεσμα εγκρίνεται. 25 υπέρ, 24 κατά. 132 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 131 αποσύρθηκε. 132. Την ψηφίσαμε, εγκρίθηκε. 133. Και 134 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος χρειάζεται. Ενδεχομένω να έχει απορριφθεί, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Έναρξη. Και πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 135 υπέρ. Κατά αποχές ε, έλεγχος. Και για αυτήν. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 29 ψήφους υπέρ. Η συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 147, 148 και 151 από κοινού. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, 149 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 160 και 161 από κοινού. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163, 164 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε για να είμαστε 100% βέβαιοι. Την 178 παρακαλώ ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε εγκρίνεται με μία ψήφο. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 199 μαζί με την 200 υπέρ. Κατά αποχές Ας το ελέγξουμε και αυτό. Έναρξη, παρακαλώ, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται με 7 ψήφους. Διαφορά. Η 201 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές απόλυτη. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές α, εγκρίνεται. Η 219 μαζί με την 220. 221, 222, 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2.24 υπέρ κατά Ας ξαναδούμε παρακαλώ. Σήκωσε τα χέρια γιατί είναι 2.24. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 227 υπέρ, α, καταπίπτει. Η 227. Λίμπε 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 230 και 231 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 243, υπέρ, κατά, αποχές, να επαναλάβουμε παρακαλώ, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 243, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 244 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 250 και 251 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 252 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α, να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 32. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη φοφορίες. Εγκρίθηκε. 34 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. 33 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 266 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 276 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 279 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 286 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 295 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 296 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Ωραία. Για τη 296 ηλεκτρονικά μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 31 ψήφι κατά. 297 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρο, εγκρίνεται. 298 εγκρίνεται. 299 τώρα υπέρ, κατά, αποχέ. θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 299. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες, απορρίφθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 301 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 και 308 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 309 και 310. Όχι, 309 υπέρ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 αποχές θα ελέγξουμε για τροπολογία 12 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω καλά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 30 ψήφοι κατά. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται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 Απορρίφθηκε πάντω. 30 ψήφοι κατά. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 40. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 41 υπέρ, κατά, αποχές. Για να είμαι σίγουρη θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τις ψηφοφορίες απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Γυναικών, ε. Α, να ελέγξουμε για τις 45. Καλώς, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. 20-20 απορρίπτεται. Γυναικών, ε, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γυναικών α, ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γυναικών J υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γυναικών C υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Γυναικών C. πέρας υποφορίας Εγκρίνεται. ΦΑΜ κάπα και α, Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο σχέδιο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με 46 ψήφους υπέρ και μία κατά. Συγχαρητήρια, κυρία Βέμπερ. θα συμπεριλάβουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην έκθεση ως Και τώρα. Περνάμε τώρα στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Θα ξεκινήσουμε με την συμβιβαστική H αγγλικό και είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά πηγαίνουμε στην 34. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 36. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική Άι Αγγλικό, υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. Η κυρία Χάρκινγκ Κυρία Χάρκιν, εξηγήστε μας. Εμείς σήμερα πήραμε κάποιες συστάσεις, προτάσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμού για να προσθέσουμε στις συμβιβαστικές μας. Είναι μία προσθήκη. Είναι τρεις προτάσεις μας έκαναν, δεχόμαστε τη μία. Εγώ δεν θα την υποστηρίξω, αλλά θα την αναγνώσω. Προτείνεται στα πλαίσια των εθήμων και των συνηθιών των κρατών μελών οι αιτήσει για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μπορούν να κατατεθούν από τις αρχές που διαχειρίζονται τα διαφθορωτικά ταμεία σε κάθε χώρα εφόσον οι αρχές αυτές έχουν τους ανθρώπινους πόρους και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Αυτή είναι η προσθήκη. Οπότε θα ψηφίσουμε επ' αυτής της προτάσεως. Υπάρχουν αντιρρήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αντιρρήσει, συνεπώ θα ψηφίσουμε επί του κειμένου το οποίο ανέγνωσε η κυρία Χάρκεν. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας με μία ψήφο διαφορά. Απερίφη με μία ψήφο διαφορά, κυρία Χάρκιν. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε τώρα την συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική και η αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 46, πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε. Έτσι ώστε να μην ε, μείνει κάτι αμφιλεγόμενο. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 46. Πέρας της ψηφοφορία. Απερίφθη. Το 47 έχει αποσυρθεί. Πηγαίνουμε στη συμβιβαστική Έλα, Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποκές, δεκτή. 49. Όχι λάθος λέει η πρόεδρος. 51. Ποιοι είναι υπέρ. 51. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική M υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ίντα 11 στη σελίδα 8. Ίντα 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. AM ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63. Υπάρχει, είναι προφορική, υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ποιοι είναι υπέρ της 63 κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 65, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 9 ψήφι διαφορά. Προϋπολογισμός 16. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική όου υπέρ, κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική Q στη σελίδα 10. Αλλά κάτι ξεχάσαμε λέει η Πρόεδρος. Συμβιβαστική πι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά πηγαίνουμε στην 10 συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή. 78 προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. 79. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική S. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στη συμβιβαστική T στη σελίδα 13. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Ρέτζι 20 Λοιπόν, Ρέτζι 20. Α, έχει καταπέσει και αυτή, διορθώνει η πρόεδρος. 93. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, δεκτή. 94 και 95. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, απερίφη. Συμβιβαστική U, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική V. ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική W, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 100, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές απερίφη. Προϋπολογισμός 7. Πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα της 7 προϋπολογισμός. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτό. Συμβιβαστική X. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. 107. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απερίφθη. 108. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απερίφθη. Συμβιβαστική Y. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Συμβιβαστική Z, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Τροπολογία 116, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 116, ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Συμβιβαστική, α όχι λάθος, τροπολογία 117. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Δεν σας βλέπω καλά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί πολλοί από εσά δεν σηκώνουν το χέρι τους. Πέρα στις ψηφοφορίες, Αυτό ήταν ένα ισχυρό ε, μήνυμα, αλλά δεν φάνηκε από τα χέρια σας. Λοιπόν, AA, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, αδεκτοί. Συμβιβαστική AB, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτοί. 127, ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Συμβιβαστική AC, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. 132, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Συμβιβαστική AD, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. 138. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 138 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική ΑΕ Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Ρέτζι 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απερίφθη. Ρέτζι 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική AF. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική AG. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 150. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. 151. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. 152. Υπέρ, κατά, αποχές. Ίσως να απορρίφθηκε, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1.52. Τέλος απερίφθη με δύο ψήφους διαφορά. AH υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 156 υπέρ κατά αποχές Η περηφάνεια μου δυστυχώς μου ζητά να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 156 λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας και απερίφθη. Με 11 ψήφους διαφορά. 157. 157 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. 158 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AI, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AJ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. ΦΑΜ 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη ΦΑΜ 10 Τέλος, δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική AK υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την AK. Άρχεται η τέλος μάλλον της ψηφοφορίας, λέει η πρόεδρος. Δεκτή. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική A. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική B. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή Συμβιβαστική AL υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ B υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφη Συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Φεμ A υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φαμ B υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Φαμ B. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή με δύο ψήφους διαφορά. Φάμψη υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτή, όπως η προηγούμενη. Ή μάλλον θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη ΦΑΜΣΥ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας με δύο ψήφους διαφορά γίνεται δεκτή. Και έχουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος όπως τροπολογήθηκε η ηλεκτρονική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. «48 υπέρ 0 κατά». Συγχαρητήρια στη Μάριον Χάκεν για την έκθεσή της. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ενσωματωθεί στο περιεχόμενο της έκθεσης. Αυτό σημαίνει <coughs> ότι περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Και αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τη σχετική οδηγία του κ. Μπαχ. Και ξεκινάμε με τη συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Συμβαστική C. Συμβαστική C πρώτα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές απορρεπτεται. Ιωνέα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21. Στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 21, παρακαλώ. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Have you all voted? Yes. παρακαλώ όλοι. Πέρα Πολύ ωραία. 24 ε, και 38 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Age ήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολογία 45, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48. Προφορική ερώτηση. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Πέρασε. Κάτι δεν πάει καλά, λέει η πρόεδρος. Κάποιο πρόβλημα? We have to repeat it. Να επαναλάβουμε παρακαλώ την ψηφοφορία της τροπολογίας 48. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι οριακό. Το βλέπετε στις οθόνες. Συμβιβαστική ΆΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πεντεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 έχουμε ένα αίτημα του Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να υποστηριχθεί από τον κύριο Μπάχ να γίνει ψηφοφορία σε μέρη. Το τελευταίο μέρος της τροπολογίας 58, το οποίο είναι το εξής. Θεωρεί ότι είναι καθήκον των εργαδοτών να δίνουν σωστή απασχόληση και να δίνουν νέες τεχνολογίες όπως ε, εφαρμογές IT και τονίζει σε περίπτωση προσωρινών συμβολέων η υπηρεσία που δίνει το προσωπικό θα πρέπει να παρέχει τη σωστή κατάρτιση και προετοιμασία. Αν εγκριθεί λοιπόν αυτό, αν εγκριθούν αυτές οι προτάσεις, θα προσθεθεί αυτό το κομμάτι στην συμβαστική ΆΗ στο τέλος. Συμφωνείτε με την ε, τμηματική αυτή ψηφοφορία. Μάλιστα. Άρα θα το ψηφίσουμε, λέει η Πρόεδρος. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε παρακαλώ την 61. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Την 61, ναι. Και τώρα λοιπόν κλείνει. Η διαδικασία της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έλεγχος δείτε για την 82. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 υπέρ 22 κατά. Ισοψηφία απορρίπτεται. Η 83 υπέρ κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική μη υπέρ κατά. Αποχές έγκρινεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολό του σχεδίου γνωμοδότηση όπω τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη τη ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ε, θα τροποποιηθεί και θα υποβληθεί αυτό στην ε, έκθεση. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπαχ. Και τώρα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διατάξη μετά την ε, ψηφοφορία. για την ε, διάσκεψη των τριών ημερών για την ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα. Μάλιστα, θα σας δώσουμε ένα λεπτό για να αποχωρήσετε ήσυχος όσοι δεν θέλουν να ακούσουν τον κύριο Σόγκορ. συνεχίζουμε με αυτό το νέο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, που είναι η τριμερής διάσκεψη για την απασχόληση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόγο, στον εισηγητή. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Σε από το 2003 διάσκεψη αυτή, σε υψηλό επίπεδο, άτυπες συναντήσεις μεταξύ Επιτροπής, Προεδρίας και Κοινωνικών Εταίρων. Ήδη από το 1997, στα πλαίσια της στρατηγικής για την απασχόληση και της στρατηγικής για τη Λισαβόνα και της στρατηγικής για το 2020. Από το 2003 όμως πρόκειται για ειδική συνάντηση στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου στο υψηλότερο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Κοινωνικών Εταίρων. Από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα, η Προεδρία του Συμβουλίου και η Προεδρία τη Επιτροπή από κοινού προεδρεύουν τη διάσκεψη αυτή. Όμω, η συνθήκη τη Λισαβόνα προχώρησε σε θεσμικέ αλλαγέ. Η μία είναι ότι δημιούργησε το ρόλο ε, της ε, προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η αναγνωρίστηκε η διάσκεψη αυτή σαν μια διάσκεψη που συνεισφέρει στον κοινωνικό διάλογο. Επίσης, η συνθήκη της Λισαβόνας επαναλαμβάνει την ίδια μορφή του άρθρου 220. Όλες αυτές οι αλλαγές χρειάστηκαν για να αλλάξει η νομική πράξη πάνω στην οποία βασιζόταν η διάσκεψη αυτή. Το TSS λοιπόν λειτουργούσε χωρίς νομική βάση από την ε, έναρξη τη ηθίκη τη Λισαβόνα. Τα κύρια στοιχεία που θα αλλάξουν τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου είναι τα εξή. Πρώτον, η νομική βάση θα είναι το άρθρο 352 της Εθνικής Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή επίσης θα αλλάξει γιατί θα αναφέρεται τώρα στρατηγική 2020 και η σύνθεση θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής, η Προεδρία του Συμβουλίου, οι δύο διαδοχικές και η κοινωνική εταίρη. Βάσει πρακτικών μέχρι τώρα, η συνάντηση γίνεται δύο φορές το χρόνο, όχι μία φορά, όπως έλεγε η απόφαση του 2003. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουμε καλά τη σημασία που έχει ο κοινωνικός διάλογος για την ε, απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας Τα ωφέλη είναι για τους εργοδότες, για τους εργοζόμενους, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση, αν θέλουμε πραγματικά οι πολιτικές μας να γίνουν κτήμα του κόσμου και να εφαρμόζονται οι αποφάσεις μας, είναι ζωτική σημασία να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι σε όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις πολιτικής. Στο μακροοικονομικό διάλογο η τριμερής ε, αυτή η διάσκεψη μπορεί να ε, βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών κάθε φορά που εφαρμόζονται πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλη σημασία οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τους Ευρωπαίους ε, ηγέτες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ήδη από τα στάδια της διαβούλευσης. Είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση αυτή, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, αναγνωρίζεται η ανάγκη για νέα απόφαση του Συμβουλίου που να λαμβάνει υπόψη το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχουμε σήμερα μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Στην τελική απόφαση υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις. Πιο συχνά γίνονται οι συναντήσεις Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει δεόντως να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των, ε, της διάσκεψης αυτής κάθε φορά που συνέρχεται. Τα πιο σημαντικά είναι ότι η πρόεδρός μας θα πρέπει μονίμου βάσεως να, να προσκαλείται στις διασκέψεις, κάτι το οποίο δεν το λέει η απόφαση του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο συμμετέχει σε πολλές αποφάσεις για κοινωνικά ζητήματα και αυτό λοιπόν είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε, να προσκαλείται η Προεδρός μας δηλαδή, αν θέλουμε αποτελεσματικό διάλογο και πλαίσιο στα κοινωνικά. Γι' αυτό προτείνω να δώσετε σύμφωνη γνώμη του το Κοινοβούλιο στην Ολομέλη για την απόφαση του Συμβουλίου, μόνο εφόσον έχουμε πάρει γραπτά επιβεβαίωση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι τρέχουσες ε, πρακτικές για την πρόσκληση του Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεχιστεί και θα επιβεβαιωθεί και στο μέλλον. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Σογκόρ. Αν κάποιος θέλει το λόγο τώρα για να αντιδράσει, να κάνει κάποια παρατήρηση, παρακαλώ, Μάιτα. Ευχαριστώ. Εδώ μιλάω για τον κύριο Μπαλάς, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, λέει ο κύριος Μαρτά. Θέλει να συμφωνήσει πάντως με τον εισηγητή, λέγοντας ότι είναι θλιβερό που το Συμβούλιο και σε ένα βαθμό και Επιτροπή όταν πρόκειται για την πρόθεση του κοινωνικού διαλόγου με τους ε, συνδικαλιστές και την εργοδοσία, δεν ε, προχωρά σε διοργανική διαβούλευση. Η τριμερής διάσκεψη δεν συμπεριλαμβάνει επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο κ. Μπάλα στηρίζει τη θέση του εισηγητή και των συντονιστών τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δώσει την τελική του έγκριση, το είπε και ο εισηγητή αυτό, στην απόφαση του Συμβουλίου, παρά μόνο αν έχει πάρει επίσημα δέσμευση από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσκαλέσει στι επόμενε διασκέψει τον πρόεδρο τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασία. Πρόεδρος. Ωραία. Άλλος. Η κυρία Χάρκιν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή και εγώ. Πράγματι πρέπει να έχουμε πρώτα την επιβεβαίωση αυτή από το Συμβούλιο, ότι όντως θα είναι συνήθις πρακτική να προσκαλεί το Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης στην διάσκεψη. Συμφωνώ με τον κύριο Σόγκουρ, δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος αλλιώς. Συμφωνώ, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πετήσουμε. Πρόεδρος. Ωραία, φαντάζομαι αυτά είχαμε να πούμε σήμερα για το θέμα. Στην Ολομέλεια θα προχωρήσουμε το Σεπτέμβριο 2016. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπω έχουμε εδώ πέρα κάποιον που θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις παρατηρήσεις σας. Το θέμα συζητιέται αυτή την εποχή και θα ενημερώσουμε. Όταν ληφθεί απόφαση θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε η απόφασή μας να είναι ικανοποιητική για σας. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Οι τροπολογίες θα είναι παραδεκτές μόνο εφόσον ανατρέπουν την προτινόμενη σύσταση έτσι όπως προτείνεται από τον εισηγητή. Όπως είπα και νωρίτερα, στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο θα έρθει το θέμα, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι το σημείο μας αριθμός 12. Νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων. Το λόγο έχει η κυρία Τζεντίλε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι η συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας για τα ζητήματα αυτά, τα οποία θίγει η Επιτροπή μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να θίξουμε το σημαντικό αυτό σημείο σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά ε, την καινοτομική αυτή διάσταση του νέου μοντέλου. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα της απασχόλησης στα πλαίσια μιας πιο ε, ευθύους ε, προσέγγισης η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες και στη ζήτηση. στη ζήτηση από πλευρά των ε, καταναλωτών. Τώρα θέμα λοιπόν τώρα είναι το τι γίνεται με την ποιότητα σε σχέση με αυτά που προσφέρονται. σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εργασία, σε ό,τι αφορά την προστασία που συνεπάγεται αυτό. είμαι ανοιχτή σε προτάσεις για βελτίωση της πρότασης, δεδομένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζητήματος των κρατών μελών. Το σύστημα λοιπόν της οικονομίας αυτής, της συνεταιρεστικής αν θέλετε ή συνεργατικής, είναι ενδιαφέρον, προκαλεί ζήτηση στις μεταφορές, στην κινητικότητα, στην προσβασιμότητα, με διασταύρωση με το θέμα το κόστος και των μέτρων λοιπόν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα μέσο αντιπαράθεσης στην ένδια των ευκαιριών και όχι μόνο στην οικονομική ένδια. Μια κινητικότητα με προσβάσιμο κόστος στο εσωτερικό ενός οράματος το οποίο εγώ πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να θέσουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, οι ιδιωτικέ μεταφορές είναι για μας ή μπορεί και να μην είναι για μας μία δημόσια υπηρεσία και θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις και προς τους καταναλωτές και τους εργαζομένους στα πλαίσια των διοικητικών δομών όπως οι αδειοδοτήσεις όχι μόνο των μεταφορών αλλά και οι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες δίδουν εγγυήσεις και επιτρέπουν στις υπηρεσίες αυτές να λειτουργήσουν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να εντοπίσουμε τη χρησιμότητα των μέσων αυτών, σε ποιο βαθμό λειτουργούν εν παροχές ε, ενδιαμέσου και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπόκεινται και ε, φορολογικό βάρος, πίεση. Μέσα από τους διαγωνισμούς, μέσα από την κατάθεση απαιτήσεων, ετοιμάτων, καινοτομιών και στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα της φορολογίας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και κανόνες οι οποίοι θα αποτρέπουν σε ορισμένες χώρες μέλη να δημιουργηθούν δυνατότητες περαιτέρω κοινωνικού ντάμπινγκ. Συνεπώς η συζήτηση αυτή είναι ενδιαφέρουσα, η συζήτηση αυτή θα, θα, επιτρέψει να υπάρξουν και άλλες δυνατότητες αντιπαράθεσης έτσι ώστε να μην αγνοήσουμε τις δυνατότητες αυτής με ποιότητα στην υπηρεσία, με ποιότητα επίσης ε, και στην μικρή επιχείρηση που πρέπει να προστατεύεται στα πλαίσια της ε, ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα νέα συνεργατικά μοντέλα πρέπει να μας προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Θέλω να υπάρξει μια συζήτηση ειλικρινής, ανοιχτή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να εμβαθύνουμε αυτό το σημαντικό κατεμέ θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σούλτς από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Πρόεδρε, η συνάδελφο Τζεντήλε πραγματικά θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί πολλά σημεία έδειξε τα οποία με απασχολούν και τα οποία παρουσιάζονται και στην έκθεση σε... και θα έπρεπε ασφαλώς να παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την ε, οικονομία την συνεργατική σε ό,τι αφορά για τα ταξί, για παράδειγμα, για τα λεωφορεία, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Παρέχουν ευκαιρίες για νέα, για νέα, για νέες θέσεις απασχόλησης. Κυρίως σε ό,τι αφορά το ταξί. Δεν έχουμε το θέμα ότι δεν αρκούν οι άδειε. Και αυτό κάνει και πιο ακριβό το να έχει κανεί συνταξή Και θεωρώ ότι αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία οι νέε τεχνολογικέ εξελίξει για να δημιουργηθεί ε, θέση εργασία. Ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν χαμηλές ε, χαμηλά προσόντα, χαμηλά επίπεδα εξειδικευσή, αλλά και για τους ε, και του πρόσφυγε μπορεί να ξεκινήσει για κανένα παράδειγμα άμεσα να δουλεύει, αρκεί να έχει ε, ένα smartphone και μόνο. Και είναι εύκολο και άμεση η χρήση των εφαρμογών αυτών. Αυτό που επίσης ε, αναφέρει η έκθεση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και περιορισμένοι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά υπηρεσίες ε, μεταφορών. Ιδιαίτερα για απομακρυσμένε ε, περιοχέ όπου δεν υπάρχουν πολλέ δυνατότητε ε, μέσων συγκοινωνία. Πιο πολλοί έχουν ε, δίπλωμα οδήγηση ή μπορούν να το αποκτήσουν αυτό σχετικά εύκολα και μπορούν λοιπόν να ξεκινήσουν γρήγορα τη δουλειά τους και δεν χρειάζεται επίσης κανείς να ξέρει καν το μέρος στο οποίο βρίσκεται γιατί υπάρχουν τα συστήματα πλοήγησης και αυτό βοηθάει ιδιαίτερα για τη μείωση της ανεργίας μεταξύ των ε, ατόμων χαμηλής εξειδικευσής και εκπαίδευσης, γιατί θεωρώ λοιπόν ότι οι ευκαιρίες αυτές είναι αυξημένες στον τομέα των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό, την ψηφιακή καμπή στον τομέα των μεταφορών, χρειαζόμαστε πιο πολύ ευελιξία στον τόπο και στον χρόνο εργασίας και προσαρμογής σε διάφορες ε, φάσεις της ζωής. Ε, μιλάμε για μικρές ε, επιχειρήσεις σήμερα και πίσω από αυτές κρύβονται συχνά αυτό Έτσι λοιπόν η συνεργατική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες Μορφέ απασχόληση. Πιστεύω λοιπόν ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών αυτών μοντέλων είναι θετική. Αλλά είναι ασφαλώ σημαντικό να τηρούνται οι νομοθεσίε. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα κοινωνικά μοντέλα, τα οποία δεν θα πρέπει να διαβρώνονται. και θα πρέπει να τονίζετε αυτό καλύτερα από ό,τι τώρα. Στην έκθεση θα ήθελα επίσης να επισημάνω δύο-τρία σημεία κριτικής. Στην παραγραφό 3, σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τις επισφαλείς ε, τρόπους απασχόλησης, να το συζητήσουμε τι ακριβώς εννοείται. Και προβληματικό είναι επίσης ε, το θέμα της εισαγωγής συνολικής ευθύνη για την ε, ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών. Θα υποβάλουμε λοιπόν τις σχετικές τροπολογίες και θα τις συζητήσουμε ασφαλώς και με την συγκεκριά. Thank you, Paloma Lopez. Σας, σας Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λόπες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Τζεντίλε, για τη γνωμοδότησή της, η οποία πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τη στιγμή που εγκαθίστεται στις μεταφορές μια επιχείρηση, πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτήν όλες οι προδιαγραφές που ισχύουν στον κλάδο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί με κόλπα συνεργατικές ε, μεθόδους όπως είναι η Uber και έτσι να υπονομεύει τους ταξιτζίδες. Τι είναι αυτή τελικά, είναι αυτόνομη, είναι μισθωτή. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση συγκεκριμένη για έναν τομέα και άπαξ και υπάρχει πρέπει να εφαρμόσετε σε όλους τους σχετικούς φορείς. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί σαν άλοθη μία ψηφιακή πλατφόρμα. Έπειτα το κοινωνικό dumping, το να διαδίδονται έτσι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις αυτόνομες στις μεταφορές, όπως είναι τα φορτηγά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρύβονται οι σχέσεις εξάρτησης και δεν πρέπει να εποφελούνται και να κάνουν κατάχρηση μία αγορά τη οποία η κατάσταση όλο και χειροτερεύει. Η ψηφιοποίηση μπορεί να οδηγήσει βέβαια στον εξυγχρονισμό και να βελτιώσει τον κλάδο, αλλά τα δικαιώματα των εργαζομένων στι μεταφορές πρέπει να είναι αυτά τα οποία υπερισχύουν ανα πάσα στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λοτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του κύριου Σορτόφσκι, θα ήθελα να πω δύο λόγια στην κυρία Τζεντήλε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το πιο δυναμικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πάνω από 30% των εργαζόμενων απασχολούνται ακριβώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεταφορές λοιπόν είναι ένας ιδιαίτερος τομέας. Στους σιδηροδρόμου και στις αερομεταφορέ υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρόσφατα, τα πρόσφατα χρόνια είδαμε ότι η δημιουργικότητα, το επιχειρήν, βοηθάει να έρθουν εμπόδια και να δημιουργηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα συγκεράζοντας παραδοσιακά μοντέλα μεταφορών με νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά δηλαδή την παραγγελία ή τις πληρωμές. Το πιο επίμαχο ζήτημα βέβαια έχει να κάνει με τις οδικές μεταφορές. Τα νέα μοντέλα επηρεάζουν την αγορά εργασίας και τις συνθήκες εργασίας. Ο κύριος Ροτοφσκή λοιπόν πιστεύει ότι η γνωμοδότησή μας θα πρέπει εντελώ ειλικρινά να αντιμετωπίζει και τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους των νέων αυτών μοντέλων. Για πολλούς νέους υπάρχουν νέες προοπτικές απασχόλησης. Προσφέρονται ευέλικτες ώρες εργασίας. Παρόλα αυτά, ελοχεύουν και κίνδυνοι. διότι πολλοί ε, πάροχοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αναλογικές ε, τεχνολογίες. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το βάρος της γραφειοκρατίας. Όσο πάντως κάποιος στηρεί το νόμο, μπορεί να δουλεύει κιόλα. Η νέα αγορά λοιπόν δεν πρέπει να περιορίζει τους εργαζόμενους στα δικαιώματά τους. Ο κύριος ε, Ζητόσκι θέλει να βρεθεί μια καλή ισορροπία, ε, μια τέτοια διατύπωση που να μην προχωράει σε διακρίσεις κατά των εργαζόμενων, ούτε κατά των επιχειρήσεων και ούτε βέβαια κατά των καταναλωτών. Θα υπάρξουν τροπολογίες που θα υποβληθούν προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, την εισηγητρία για την γνωμοδότηση. Περιλαμβάνει πάρα πολύ καλέ ιδέε και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία μαζί της. Από πλευρά. μου. Ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν καινούριο τομέα και υπάρχουν τόσο πολλοί άγνωστοι παραγοντέ. Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι πολύ κατακριματισμένο στην παρούσα φάση και πολλά διαφορετικά σημαίνουν στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη πρόκληση να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτά που ανέφερε και η προηγούμενο ομιλητή. Μία ισορροπία μεταξύ του καταναλωτή, του εργαζόμενου και των υπηρεσιών που παρέχονται. Από αυτή την άποψη λοιπόν πιστεύω ότι ξεκινάμε ένα ολόκληρο ταξίδι αν θέλετε και προφανώς υπάρχουν ε, ωφέλη σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες και μεγάλες δυνατότητες για την απασχόληση. Έχουμε τη δυνατότητα για ε, ευέλικτα ωράρια εργασίας ε, και για όσους το επιθυμούν αυτό είναι πολύ θετικό γιατί αυτό αποτελεί μια νέα πηγή εισοδημάτων. Θα συζητάμε και θέματα, θα συζητήσουμε και θέματα ισορροπίας ιδιωτική και επαγγελματική ζωή και προφανώ η συνεργατική αυτή οικονομία έχει σημαντικό ρόλο να παίξει προ την κατεύθυνση αυτή. Θα παρέχονται και νέε υπηρεσίε, θα υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμό. Και υπάρχει σίγουρα πρόκληση σε ό,τι αφορά του υφιστάμενου φορεί και παράγοντε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιον τρόπο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισότητα σε ό,τι αφορά την συνεργατική οικονομία. θέτει τις προτεραιότητες ό,τι αφορά την, τα περιουσιακά στοιχεία. Σε όλα αυτά λοιπόν είναι θετικά στοιχεία. Και νομίζω ότι πολλά πολλά ζητήματα έχουν σχετίζονται με την ε, νομοθεσία. Το τι λείπει, το τι περιλαμβάνεται, πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Γιατί προφανώς ε, δεν είναι σαφή τα πράγματα ε, μεταξύ των εργαζομένων, των καταναλωτών, των παρόχων, των αυτοαπασχολουμένων και όπως σα είπα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και θα τα συζητήσουμε επί μακρόν. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ε, νομικές αμφιβολίες για τους ορισμού σε ό,τι αφορά τον πάροχο υπηρεσιών, τον ενδιάμεσο για παράδειγμα και νομίζω ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αβεβαιότητες, αυτό μπορεί να αποτρέψει τον ε, σωστό και ίσο Η συνεργατική επιχείρηση είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα από διαφορετική προοπτική. Κάπου πρόσφατα διάβαζα, εντάξει δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή η ιδέα και στον τουρισμό και τα τρόφιμα είναι το θέμα του, των τροφίμων που μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Δεν ξέρω τα εστιατόρια πώς θα το χειριστούν αυτό. Να είμαστε πάντως προσεκτικοί ε, για να μην υπάρχουν και ε, ανταγωνισμοί σε αυτά και για τις προτάσεις του εισηγητού να μην υπάρχει φοροαποφυγή, συμφωνώ, και να υπάρχουν και σαφείς ορισμοί για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Σίγουρα μπορώ να συμφωνήσω με όλα αυτά. Οπότε προσβλέπω και εγώ σε παρεντέρω συνεργασία με την εισηγητρία. Σε ευχαριστούμε, Λαώρα Άγκια τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Τίλε για την πρότασή της στα πλαίσια της διατύπωσής της υπάρχουν στοιχεία με τα οποία εμείς θα συμφωνήσουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες παρατηρήσεις από πλευράς μας, γιατί σήμερα η τεχνολογική πρόοδος στα πλαίσια αυτής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς δεν είναι σε θέση να προσδώσει αυτή την προστιθέμενη αξία την οποία επιθυμούμε, γιατί δεν υπάρχουν οι κοινέ βάσεις στις διάφορες χώρες, γιατί νομίζω ότι αν δεν προσέξουμε θα αυξήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εφόσον θέλουμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την ενιαία ψηφιακή αγορά, απαιτούνται κοινά σημεία εκκίνησης. Πολύ συχνά οι τεχνολογικές διαδικασίες, η ψηφιοποίηση είναι κατά κάποιο τρόπο ε, βήματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν και αρνητικές καταστάσεις γιατί στα πλαίσια της τεχνολογίας ε, δεν συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές γνώσεις αν θέλετε και υπάρχει μια θα έλεγα απομάκρυνση από την τεχνολογική στήριξη και απώλεια εμπειρογνωμοσύνης. Συνεπώς θα συμφωνήσουμε με τη συνάδελφο Τζεντίλε ε, σε σχέση με το σημείο 4. Αναφέρεται η κυρία Τζεντίλε στην υπόγεια εργασία, στο κοινωνικό ντάμπινγκ, στη μαύρη εργασία, και στην αβέβαιη μορφή απασχόλησης ε, προβλήματα τα οποία φύγουν κυρίως στις μικρομεσαίες. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει ακραία διαφάνεια σε σχέση με τους διαγωνισμούς και τις δημόσιες προμήθειες μέσω υπεργολαβιών γιατί πολλές φορές έτσι ανοίγει ο δρόμος σε απαράδεκτες συμπεριφορές σε αθέμητες συμπεριφορές Θα συμφωνήσουμε επίσης όταν μιλάτε για το σεβασμό του ωραρίου εργασίας και θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά εδώ στα πιθανά μέσα για την παρακολούθηση ας πούμε της στήρησης του ωραρίου εργασίας και του ωραρίου ανά, ανάπαυσης, να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του καμποτάζ μέσω των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμβατότητα και να υπάρχει μια σωστή θα έλεγα μορφή συνδυασμού ανάμεσα στην εργασιακή πλευρά της ζωής και στην ιδιωτική. Πρέπει επίσης να υπάρξει αναφορά και ε, σε ό,τι έχει σχέση με την υγεία των εργαζομένων στον επαγγελματικό χώρο. Ε, θα έλεγα έχουμε πολλά εδώ να δούμε και γι' αυτό θα ήταν σωστό να ζητήσουμε την σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων. Συνεπώς λοιπόν ευχαριστώ για μία ακόμη φορά την κυρία Τζεντίλε. Είναι καλή η βάση συζήτησης που προτείνει. Ευχαριστώ κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αναφερόμαστε στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις μεταφορών. Δεν μιλάμε για τις α, ε, α, ε, θαλάσσιες μεταφορές, δεν μιλάμε ε, για τις εναέριες μεταφορές. Μιλάμε για τα ταξί ας πούμε. Μιλάμε για τους μεταφορείς δεμάτων και για το καμποτάζ, όπως επίσης και στην παραποτάμια μετακίνηση ε, προϊόντων. Στη Γαλλία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιες τέτοιες μικρές δραστηριότητες ε, μπορούσαν να ανταμείψουν αυτούς που εργαζόντουσαν σκληρά. Υφίστανται όμως ε, την λεγόμενη ουμπεροποίηση των συνθήκων ε, εργασίας και δραστηριότητας και μέσω ακριβώς του αθέμητου ανταγωνισμού Νομίζω ότι έχουν ανάγκη να εργαστούν, δεν υπόκεινται στους ίδιους φορολογικούς και οικονομικούς κανόνες από ό,τι στο παρελθόν και γι' αυτό αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πολύ στην πρόταση Gentile είναι τα σημεία 3, 4 και 5 όπου ε, τίθεται το θέμα της ε, ε, εφαρμογής των ιδίων κανόνων και κοινωνικών και εργασιακών και οικονομικών. Θα συνεργαστούμε μαζί σας με χαρά, ε, κυρία Τζεντήλε. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 27 Ιουνίου. Ε, εξέταση τροπολογιών 31 Αυγούστου και θα ψηφιστούν στην Επιτροπή μας στις 26 Σεπτεμβρίου στην κυρίαρχη επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιασλοβιέλκα που είχε ζητήσει ε, προηγουμένως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει προηγουμένως στην Επιτροπή, αλλά το οποίο νομίζω ότι θα ε, προκαλέσει ενδιαφέρον στο μέλλον και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλές εκθέσεις δημιουργείται μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας οι νέες μορφές ε, απασχόλησης γίνονται αντικείμενο συζήτησης και περιγραφής. Στην δική μας Επιτροπή εμείς δεν συζητάμε πάρα πολύ για αυτές τις νέες αν θέλετε μορφές εργασίας και για τις νέες δυνατότητες και γνώσεις που απαιτούνται. Η κυρία Χάρκινγκ είπε ότι τα φαινόμενα αυτά βρίσκονται σε παιδική ηλικία, αλλά η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με τρομερή ταχύτητα και θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Και η κυρία Ατζία αναφέρθηκε επίσης στην διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες επαναστατικές αλλαγές να συμβαίνουν και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτριά μας έτσι ώστε στις δικές μας ε, επιτροπές να φωνάξουμε και εμπειρογνώμονες να μας μιλήσουν για το τι αλλάζει, για το τι συμβαίνει. Η Μάριον αναφέρθηκε στις εξελίξεις σαν παράδειγμα στον τουρισμό. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με το μέλλον των επιχειρήσεων ε, και το μέλλον των μικρομεσαίων είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς ε, ε, να αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να στρουθοκαμιλίζουμε, πρέπει ε, να ανταλάβουμε υπόψη μας. Συνεπώς λοιπόν να φωνάξουμε εμπειρογνώμονες για να μας μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Ουλσκόγκ για την παρέμβασή σας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συντονιστές καταρχάς να κάνουμε πράγματι συναντήσεις και να προσκαλέσουμε ανθρώπους που έχουν γνώσεις γύρω από αυτά και πρακτικές εμπειρίες. Εμείς τα θέματα αυτά μας ενδιαφέρουν, αλλά δεν ε, μας ενδιαφέρουν με τόσο οργανωμένο τρόπο όσο θα έπρεπε. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρότασή σας. Αυτό ε, Έκλεισε το θέμα λοιπόν με την κυρία Τζεντίλε. Τώρα θα ξεκινήσουμε το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις ε, πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Η κυρία Ατζέα είναι η υπεύθυνη και της δίδω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη ε, δύναμε. Πήρα τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες και από τους σκιώδεις. Τους ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο το να συνεργαστούμε στενότερα. Έχω προετοιμάσει ήδη ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίε ελπίζω θα αντικατοπτρίζουν τις τάσεις οι οποίες επικρατούν στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές έχουν ε, τηρούν στάση κριτική σε σχέση με την λεγόμενη στρατηγική 2020. Ε, Οι στόχοι φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την δυνατότητα που είχαμε να τους πετύχουμε πρόσφατα και νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε χαίνοντα προβλήματα όπως τη μακροπρόθεσμη ανεργία, όπως την ανεργία των νέων, όπως την δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για την αντιμετώπιση της φτώχειας των παιδιών, γιατί φύγει η φτώχεια αυτή τις παιδικές ηλικίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα, πώς θα μπορέσουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το θέμα του διαλόγου με, τις, με τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους. Ε, έχουν κατατεθεί και ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα άρθρα η γραμματεία μας είχε ήδη βέβαια ζητήσει να μην δράσουμε πάνω στα μεμονωμένα άρθρα, αλλά να περιοριστούμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Πάντως, στα πλαίσια των συναντήσεων που ε, είχαμε και με τους ε, νομομαθείς του Κοινοβουλίου θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει η πρόταση ας πούμε της σοσιαλιστικής ομάδας για το κομμάτι του κειμένου το οποίο επαναλαμβάνει τις θέσεις που δημοσίευσε και υιοθέτησε βέβαια πρώτα το Κοινοβούλιο πέρυσι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή ή μήπως θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μια ενιαία συμβιβαστική πρόταση για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις ε, ρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ ακόμα για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια της, ε, των συναντήσεων των σκιωδών. Θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ για τους σκιώδεις. Παρακαλώ. Ε, κυρία Ιασλόφιτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά. Και εκ του ΕΛΚ θα ήθελα να εξηγήσω κάποιες από τις τροπολογίες που προτείνουμε, για τη 13 για παράδειγμα, η οποία ζητάει περισσότερη συμμετοχή των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής μας για το 2020. Η τροπολογία 20 επίσης αναφέρεται στη σημασία που έχει το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης που δημοσιεύτηκαν το 2015 δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο επαρκώς και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Τροπολογία 25. Αυτή αναφέρεται στη συμφωνία όσον αφορά την έκθεση Ριμπέρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Επιτροπή μας πρέπει να ζητάει τρεις δείκτες απασχόληση για την νεολαία, μακροχρόνια ε, αναργία. Δείκτες οι οποίοι να παρακολουθούνται κάθε φορά. 33. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία απασχόλησης και σε μια δυναμική αγορά εργασίας με τη συμμετοχή όλων. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στις τροπολογίες του Σβέν Σούλτσε που στηρίζουμε. Τροπολογίες 9, 10, 14, 22, 23, 25, 28 και 31. Αυτές οι τροπολογίες είναι προβληματικές για την ομάδα μας γιατί έχουν να κάνουν με τη λιτότητα, αμφισβητούν ε, την αξία των κατευθυντηρίων γραμμών και αναφέρονται σε κοινωνικούς δείκτες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τους σοσιαλιστές να εξηγήσουν την τροπολογία 39. Και τι γίνεται με τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015. Θα πάρει υπόψη το Συμβούλιο την άποψή μας. Εγώ δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θα εκτιμήσουν να συμπεριλάβουμε αυτό το copy-paste στη γνωμοδότηση αυτή είναι σαν να έχουμε λίγη φαντασία. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ε, περισσότερο συζήτηση για το τι χρειαζόμαστε βραχυπρόθεσμα και τι μπορούμε να αφήσουμε για αργότερα, ώστε οι χώρες μέλη να κάνουν και τα αναγκαία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αβιλόπες από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αγία. Έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες περιπτώσεις και θα σας εξηγήσω ποια είναι η δικιά μας ανάλυση για το θέμα και γιατί έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και ποιος είναι ο στόχο μας. Λοιπόν, πρώτον, δυστυχώ, δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Εμείς αντιδρούμε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεχίζει στην ίδια γραμμή και για την κοινοβουλευτική μας επιτροπή έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς λέμε λοιπόν τι πολιτικές απασχόλησεις θα έπρεπε να υλοποιηθούν, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια δεν μας άκουσε, δεν άκουσε τις προτάσεις μας. Μας παρέκαμψε πέρυσι. Φέτος λοιπόν θέτουμε το ίδιο ζήτημα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ακριβώς τις ίδιες προτάσεις που υπέβαλε και πέρυσι. Θεσμικά μιλώντας, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε να καταδείξουμε ότι δεν πρέπει την θέση μας να την παίρνουν έτσι τόσο πρόχειρα. Βέβαια το Συμβούλιο θα πάρει την τελική απόφαση, αλλά δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αγνοεί, να έχουμε δουλέψει με συγητές, με σκιώδες συγητές, ε, Πυρογνώμονε και μετά όταν έρθει η στιγμή της αλήθειας για τις αποφάσεις, που σίγουρα το Συμβούλιο θα τις πάρει, τελικά να μην μας λαμβάνουν υπόψη, να μην λαμβάνουν καν υπόψη τη θέση μας. Αυτή είναι η αρχική μας λοιπόν τοποθέτηση. Θεσμικά ε, είναι πιο πολύ το ζήτημα, δεν είναι τόσο ιδεολογικό, είναι θεσμικό. Θελήσαμε λοιπόν να υποβάλουμε τροπολογίες προς διάφορες κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε αυτό που έχουμε πει, που δεν είναι και λίγο, να υποστηρίξουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και κυρίως το κείμενο που εγκρίναμε το 2015. Δεύτερον, θέλουμε να μιλήσουμε για τους στόχους της στρατηγικής 2020 και όπως ακούσαμε να εξηγήσουμε ότι κάθε μέρα πλησιάζουμε κάποιους στόχους κοινωνικούς ή ένδυες που μπορεί να μην είναι υποχρεωτικοί, αλλά αν μη τι άλλο θέλουμε να τους πετύχουμε ανισότητες, φτώχεια, περιθωριοποίηση, φτώχεια των παιδιών, όλα αυτά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας, την απασχόληση. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε μνήμα σε αυτά. Και το τρίτο είδος των τροπολογιών μας έχει να κάνει με το πώς οι στόχοι αυτοί θα γίνουν πιο δεσμευτικοί, υποχρεωτικοί της στρατηγικής 2020. Είπαμε, έχουμε δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, εισάγουμε λοιπόν τους κοινωνικούς δείχτες στο ευρωπαϊκό εξάμεινο που είναι ο σκληρός πυρήνας που απαιτεί κάποια εναρμόνιση. Αυτή, λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κατηγορίες των τροπολογιών μας. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις εισηγητές. Εγώ δεν λέω ότι εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε copy-paste το κείμενο, Εντάξει, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Να βρούμε μια διατύπωση με την οποία ε, να συμφωνήσει και η σκιώδηση συγγήτρια από το ΕΛΚ. Η πρόθεσή μας πάντως είναι να επενθυμίσουμε σε ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι πολλές φορές κάνουμε δουλειά και μετά δεν μας λαμβάνουν υπόψη το έργο μας αυτό, κανένας δεν το υπολογίζει. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει κείμενο το οποίο δεν έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι όταν κάνουμε μια δουλειά να το υπενθυμίζουμε ότι έχει γίνει αυτή η δουλειά, να μην το ξεχνάνε. Αλλά θα συμφωνήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές για να ξαναδούμε την γνωμοδότηση και να μπορέσουμε όλοι να την υποστηρίξουμε. Γιατί αυτό είναι και το χαρτί που μπορούμε να παίξουμε εμείς μέσα σε αυτό το θεσμικό τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκινγκ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ασχολείται με ένα ενδιαφέρον θέμα Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε, θα ήθελα όμως να πω ότι μία από τις τροπολογίες που κατέθεσα εξ ονόματος της ομάδας μας είναι ακριβώς ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου δεν ελήφθησαν υπόψη σε σχέση με ε, τις ε, πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών το 2015. Το δηλώνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα και ευχαριστώ την εισηγήτρια να το λάβει υπόψη της θα πρέπει να συζητήσουμε για την τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι ε, θα μπορέσουμε εμείς ε, να ε, κάνουμε μια κάποια ιεράρχηση αυτών των στόχων. Είναι δύσκολο μερικές φορές και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο, πιο πειθαρχικοί θα έλεγα για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε εν πάση περιπτώσει να έχουμε ένα ε, τελικό έγγραφο το οποίο να αντικατοπτρίζει τα θέματα τα οποία μα ε, μας ενδιαφέρουν κυρίως και να μην μείνουμε στις λεπτομέρειες. Έχουμε τρεις τροπολογίες ε, οι οποίες ε, έχουν ε, να υπογραμμίσουν ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πετύχουν τους στόχους του 2020 και υπάρχει και το θέμα της φτώχειας των παιδιών. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να συνεχίσουμε. Ο κύριος Σιλικιώτης. Πρόεδρε, ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Λάουρα για τη δουλειά που κάνει μέχρι τώρα να πω ότι και εμεί στο παρελθόν συνεργαστήκαμε μαζί με την Λάουρα, και είμαστε σίγουροι πω τέτοια θα είναι και τώρα η συνεργασία μα πολύ καλή. Ε, το πρώτο σημείο που θέλω έχω να πω, ότι εμεί δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την Επιτροπή. Αυτό η στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει αυτό που είπαμε πολλέ φορέ το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην Ένωση μα και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί ε, κάποιες πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε. Εκείνο που έχει σημασία όμως, εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να επιμένουμε σε κάποιες πολιτικές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχει τόση μεγάλη κρίση σε πολλές κράτη-μέλη και υπάρχουν ψηλά ποσοστά ε, ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Ε, οι, οι κύριες μας τοπολογίες ως ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς εκφράζουν πρώτα-πρώτα την ανησυχία μας αναφορικά με τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα ε, τα φτωχά εργατικά στρώματα, οδηγώντας τους βέβαια στην ενεργία, στη φτώχεια, την ανασφάλεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και βεβαίως στη διάλυση των εργασιακών ε, σχέσεων και σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που στην παράγραφο 1 ζητούμε δουλειά με δικαιώματα και την πρόθεσή του από τα κράτη-μέλη, στην παραγράφο 2 εισάγουμε τη συζήτηση τη ανάγκη οριστικών πολιτικών που θα προάγουν κυρίω τι δημόσιε επενδύσει για δημιουργία τέτοιων αξιοπροπόθεσεων θέσεων εργασία που θα ενδυναμώνουν κατά την άποψη μας και το κοινωνικό κράτο, ενώ στην παράγραφο 3 και 4 τονίζουμε την ανάγκη να ενδυναμωθούν τα κράτη-μέλη στη δημιουργία των δικών του στρατηγικών απασχόληση, βασισμένα στι δικέ του ανάγκε και προτεραιότητε γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι λάθος να θεωρούμε ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική για όλα τα μέλη από τη στιγμή που υπάρχουν και ε, ε, περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη, από τη στιγμή που σε διάφορα κράτη υπάρχουν ε, διαφορετικές προτεραιότητες και ανάγκες και για μας η θέση πρέπει να είναι μια εκ διαμέτρου αντίθεση κατεύθυνση από τα μέτρα λιτότητας, τα μνημόνια τα οποία έχουν καταστρέψει και οι οικονομίες έχουν καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό σε πάρα πολλά κράτη και έχουν οδηγήσει ε, στην ε, καταστρατήγηση συνεργασιακών δικαιωμάτων. Ε, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντα ότι εμεί προσλέπουμε σε μια καλή συνεργασία και με την Λάουρα και με του άλλου εισηγητέ, ώστε να βγάλουμε το καλύτερο ε, δυνατό και θετικό αποτέλεσμα μέσα από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε, κύριε Μαρτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση ξεκίνησαν από το 1998 και μας ε, εκπλήσει η ομοιότης όλων ε, των ε, εκδοχών που περιλαμβάνουν τους ίδιους στόχους διατυπωμένους μάλιστα με τον ίδιο τρόπο και 20 χρόνια περίπου αργότερα, το είπαν νομίζω όλοι, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Και συγχαίρω την κυρία Ατζέα για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνει με επιμονή και υπενθυμίζει το πρόβλημα ξανά και ξανά. Η ενέργεια των νέων είναι ένα εύλογο παράδειγμα. Το 2003 και το 2008 θέσαμε ως στόχο την απασχόληση ή την κατάρτιση 4 με 6 μήνες ε, μετά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Βρισκόμαστε στην ίδια αρχή. Το 2016 η ανεργία των νέων στην Ευρώπη είναι περίπου 20% και 50% σε ορισμένες χώρες μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Εξού και μπορεί κανείς να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. Μπορούμε λοιπόν να αμφισβητήσουμε, το είπανε και όλοι, το δεδομένο που θέτουμε ως ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση. Το σημείο κίνησης και ένα από αυτά, και εδώ θα διαφοροποιηθώ από τους άλλους συζητητές, είναι ότι ο ισχυρισμό ότι αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό με τη μετανάστευση και την ελεύθερη μετακίνηση, θα βελτιώσουμε την κατάσταση της απασχόλησης και τις θέσεις απασχόλησης, την ποιότητά τους. Κι όμως έχουμε φτάσει στις 21 Ιουνίου του 2016 και έχουμε πετύχει ακριβώς το ανάποδο. Οπότε, η πρόταση για τη μετανάστευση που ρητά αναφέρονται στις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές με τη, για την ε, απασχόληση δεν έχουν εξαφανιστεί φέτος. Απλώς το θέμα της μετανάστευσης ε, βάζει ένα επίστρωμα ανθρωπιστικής διάστασης. Δεν μιλάμε πια για οικονομικούς μετανάστες, μιλάμε για πρόσφυγες, πολιτικούς πρόσφυγες μάλιστα. Ο Άλμπερ Αϊνστάιν έλεγε ότι ο ορισμός της τρέλας είναι να ξανακάνουμε πολλές φορές το ίδιο πράγμα, ελπίζοντας κάθε φορά ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, παρόλο που επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο είναι σωστές οι ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι να συνεχίζουμε να κάνουμε τέτοια λάθη ξανά και ξανά. Και ευχαριστώ τους άλλους συνεισηγητές οι οποίοι δέχονται να συζητήσουμε και πάλι για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μας και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. 13 με 14 Ιουλίου θα ψηφίσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτήν την ε, συνεδρίαση, η οποία κράτησε τελικά πολύ. Και θα τα ξαναπούμε πριν ε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 13 Ιουλίου και στις 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. And thank you to the translators. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος που ήσασταν εδώ μέχρι τώρα.